Καλησπέρα σας. If you... I think we Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, καθότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 6 ακριβώς, όπως είπε και η πρόεδρος σήμερα το πρωί. Στην αρχή λοιπόν της δεύτερης αυτής της συνεδρίασης χαίρομαι που μπορώ να δώσω κατευθείαν το λόγο στην κυρία Μαγκίνης, η οποία είναι αντιπρόεδρος, διαμεσολάβρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις απαγωγές παιδιών από Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι που είστε εδώ σήμερα και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία του ρόλου του οποίου μόλις ανέλαβα ως διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι Απαγωγέ παιδιών. Σα παρακαλώ, με ακούτε, γιατί έχει φασαρία. Να σας παρουσιάσω λοιπόν ποιε είναι οι εμπειρίες μου και οι απόψεις μου στα εισαγωγικά μου σχόλια, εν συντομία, γιατί έχουμε εδώ και τους εμπεριογνώμονες που θα μας παρουσιάσουν τη μελέτη αυτή. Να, σε, να σας συγχαρώ όσοι ξεκινήσατε την δουλειά αυτή, γιατί ασφαλώς πρόκειται για ένα θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι θα ταιριάξει πολύ και με τα δικά μου καθήκοντα και με τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζοντας σημεία προβληματικά. Μίλησα σήμερα σε μια τέτοια συνεδρίαση διαμεσολαβητών και αυτό που ακολουθήσαμε ως γραμμή είναι ότι πάντα ακολουθούμε το καλύτερο για το παιδί. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι διάφορες δικαιοδοσίες έχουν διαφορετική ερμηνεία για το τι είναι το καλύτερο για το παιδί. Και έχουμε νομολογία για παράδειγμα που βλέπουμε δύο δικαστήρια σε διαφορετικά κράτη-μέλη να αποφαίνονται για την ίδια υπόθεση και να τοποθετούνται διαφορετικά. Αυτό είναι ένα θέμα διαφορετική ερμηνεία. Προφανώ εδώ πέρα επικρατεί η Σύμβαση τη Χάγη και η Βρυξέλλε 2. Η ιδέα είναι ότι τα παιδιά που απαγάγονται θα πρέπει να επιστρέφονται στην ε, πατρίδα τους. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Η διάρκεια αυξάνεται. Οι έξι εβδομάδε που αναφέρονται στη σήμαση της Χάγιας συχνά δεν τηρούνται. Συχνά παίρνει χρόνια και καμιά φορά ακόμα και με δικαστική απόφαση. Δεν εκτελείται η δικαστική απόφαση. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη για διαμεσολάβηση και οι σημερινέ σκέψει ήταν πολύ σημαντικέ προ την κατεύθυνση αυτή. Προφανώ, στο δικό μου γραφείο αντιμετωπίζουμε άτομα που είναι πάρα πολύ τραγμένα γιατί οποιοδήποτε έρχεται στο γραφείο μου έχει περάσει τέτοιε διαδικασίε. Και θα ήθελα να πιστεύω ότι όλα όσα κάνουμε είναι καθοδηγητικά για το κατά πόσο μπορούμε να παρέμβουμε, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, τα εκάστοτε κράτη-μέλη και να δίνουμε κατευθύνσεις και συμβουλές σε ανθρώπους που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Προφανώς πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη δυσκολία της κατάσταση και ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω μετά από κάποιους μήνες στο, στη θέση αυτή είναι να εξετάσω το πώς λειτουργεί το γραφείο. Να δούμε πώς θα πρέπει να το μετανομάσουμε. να εξηγήσουμε διαφορετικά τις ε, αρμοδιότητες τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει, θεωρώ, επισκόπηση του θέματος. Εκλεγόμαστε από διάφορα κρατημέλη για να συντονίζουμε το τι συμβαίνει στα κρατημέλη για τα θέματα αυτά. Προφανώς εξετάζουμε τις πλέον δύσκολε υποθέσεις. Είναι σημαντικό όμως να ξέρουμε ποιε είναι αυτές προκειμένου να βγουν συμπεράσματα και να γίνουν συστάσεις και αλλαγέ. Και προφανώς χρειάζονται αλλαγέ. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο το δικό μου γραφείο που δέχεται τέτοιε συστάσεις και τέτοιε υποθέσεις. Η Επιτροπή ε, Αναφορών, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και άλλα σώματα ε, στα οποία απευθύνονται οι Βλέπω και τον συνάδελφο από την Επιτροπή Αναφορών. Μπορεί να πάρει το λόγο αργότερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι όλο ένα και αυξανόμενο ο αριθμό των πολύ προβληματικών υποθέσεων και τα παιδιά υποφέρουν και, και οι γονεί, αλλά εμά μα ανησυχούν τα παιδιά βασικά. Και πρέπει να δούμε πώ θα βελτιώσουμε λοιπόν την νομοθεσία, αλλά και κυρίως την εφαρμογή. Όσο πιο μεγάλο το χρονικό διάστημα είναι που ένα παιδί έχει φύγει από την πατρίδα του, τόσο πιο δύσκολο είναι να γίνει μια αποτελεσματική επιστροφή σε αυτή την ε, πατρίδα του. Και η ζημιά που γίνεται στα παιδιά αυτά, όταν τα πράγματα έχουν ε, φτάσει στο σημείο αυτό και οι σχέσεις έχουν καταρρεύσει σε αυτό το βαθμό, είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανεί ε, τα προφανή. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη πληροφόρηση. Θέλουμε τα δικαστηρία να μπορούν να αποφαθούν τι είναι το καλύτερο, να υπάρχουν βάσει δεδομένων ενδεχομένω για να αποφασίσουμε προ τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε και σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση για το οικογενειακό δίκαιο για όλου μα προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Θα κλείσω με μία παρατηρήση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα ότι είναι πολύ σημαντική η ακρόαση και προσβλέπω και στην ανάγνωση της πλήρους έκθεσης έχω διαβάσει την αιτιολογική συστολογικές σκέψεις και την ε, περίληψη και με έχει βοηθήσει. Είναι πολύ καινούριο αυτό το τομέα εργασία μου στο Κοινοβούλιο και εγώ προσωπικά πρέπει να σα πω ότι με απασχολεί το θέμα αυτό, αλλά και πολιτικός με ενδιαφέρει το θέμα. Τα δικαιώματα των παιδιών και οι ζωέ των παιδιών είναι πολύ σημαντικά και όταν δέχονται τέτοιε βλάβε τόσο νωρί τη ζωή του, σίγουρα θα υπάρχουν ε, επιπτώσει. Και λοιπόν το δίκαιο θα πρέπει, η νομοθεσία θα πρέπει να συνδράμει στι οικογένειε αυτέ τι δύσκολε καταστάσει. Η συνθήκη τη Χάγη, την οποία υποταχθήκαμε μόλι 8 καινούριε χώρε, σα είπα στην παρουσίασή μου ότι είναι σαφή η συνθήκη της Χάγης και οι νομικές διδάξεις. Δεν είναι η πράξη όμως τόσο σαφής. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Δεν τηρούνται οι προθεσμίες. Υπάρχει σύγχυση μεταξύ των μελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σα εύχομαι λοιπόν ε, καλέ εργασίε και προσβλέπουμε στην παρουσίαση τη μελέτη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν κυρία Μακίνε, λέει η πρόεδρο. Μα πείσατε, μας πείσατε, είστε πολύ πιστικοί. Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση της μελέτης από πλευράς του κυρίου Πρετέλη από το Ελβετικό Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου στη Λοζάνη. Κύριε Πετρέλη, Πρετέλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, είναι φορτισμένο συστηματικά αυτό το θέμα και φάνηκε και από την ε, μελέτη μας. Θα δώσω όμω τον ε, Jack Current, ε, τον συνέλφο το λόγο, να σα πει τα στατιστικά στοιχεία τα οποία εκείνο είχε χειριστεί. Good afternoon. Καλησπέρα σα. Στα πλαίσια αυτή τη μελέτη συγκεντρώσαμε κάποια δεδομένα, πληροφορίε για απαγωγέ ε, των παιδιών με τη βάση διασυνοριακών γάμων και διαζυγίων. Τα στοιχεία θα βγουν συλλεγεί από δικαστικέ, ποιοκτικέ αρχέ. Δεν είναι βέβαια το σύνολο του τοπίου. Ενδεικτικά. Ξεκινάμε το 2008. Και ανατρέχουμε το 2007 και φτάνουμε μέχρι το 2012. Σε εθνικό επίπεδο η κάθε χώρα έχει κάποια στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε συγκριτικά. Να δούμε πρώτα πρώτα γάμοι και διαζύγια. Διασυνοριακή γάμοι επομένω ή ε, γάμοι δύο ε, ξένων που ζουν στην ίδια τρίτη χώρα. Δεν έχουμε πάντοτε όμως τέτοια συλλογή από, από όλα τα κράτη και το πάντως από αυτά που προκύπτουν τώρα λέμε ότι στις περισσότερες χώρες είναι σταθερό ο ρυθμό των διασυνοριακών διεθνών γάμων. Πρώτα απ' όλα λέμε ότι υπάρχει μια σταθερή άνοδος και κατόπιν πτώση όσον αφορά το, το ποσοστό στις διεθνείς γάμους και μετά βλέπουμε ότι αυτό έχει, έχει πέσει το ποσοστό αλλά πάντως σε κάθε χώρα η εξέλιξη της καμπύλης είναι διαφορετική αντίθετα σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε όλα τα δεδομένα η αναλογία των διεθνών ε, διαζυγίων έχει αυξηθεί κατά την ίδια περίοδο και έχουμε κάποια στοιχεία το 2012 και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται το, το, το 2007 ε, από το 2007 μάλλον ε, είχαμε περίπου το ίδιο ποσοστό ε, των διαζυγίων. Τώρα για να δούμε όσον αφορά τώρα την απαγωγή από τους γονείς έχουμε τη βάση δεδομένων της Σύμβασης της Φάγης της Χάγης το 2003 και 2008 έχουμε στοιχεία σε αυτή την περίοδο και επίσης έχουμε και κάποια άλλα κράτη τα οποία έχουν προσθέσει κάποια στοιχεία πιο πρόσφατα. Και ένα από τα χαρακτηριστικά της μας βοηθάει να καταλάβουμε το τι γίνεται όσον αφορά τις απαγωγές γιατί μιλάμε για στοιχεία στοιχεία 13 ετών που έχουν συλλεξεί κάποιες χώρες. Όλο και περισσότερες αιτήσει επιστροφής υποβάλλονται και η κυρία Πετρέλη ξανά έχει τη σκητάλη. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Τζον, μας μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ γιατί ήδη είπες ε, ποια είναι τα βασικά κενά όσον αφορά τη συλλογή αυτών των στατιστικών δεδομένων. Να σας πω τώρα ακριβώς ποια είναι τα κενά στο νομικό καθεστώς όσον αφορά την ε, υλοποίηση, την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης. Γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές όπως ε, προκύπτει από την ανάλυση της κατάστασης. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε τώρα τη Σύμβαση της Χάγης και τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Θα πρέπει να ενισχυθεί επομένως ο μηχανισμός ο οποίος ξεκίνησε από τη Σύμβαση της Χάγης που προβλέπει την επιστροφή του ανηλίκου στο περιβάλλον στο οποίο ζούσε πριν απαχθεί. Και επομένως ε, ε, θεωρήθηκε ότι έτσι θα υπάρχει μια ανάσχεση του φαινομένου, θα αποτραπεί η απαγωγή και θα αποθαρρυνθούν οι απαγωγείς. Όμως είδαμε ότι δεν επετεύχθη το αποτέλεσμα αυτό. Σύμφωνα με τις στατιστικές διαπιστώνουμε ότι μάλλον το αντίθετο έγινε και γι' αυτό και έχουμε τις επιστροφής πολύ περισσότερες. Για να δούμε τώρα γιατί χρεοκόπησε αυτή η προσπάθεια ανάσχεσης του φαινομένου. Θα μπορούσαμε να πούμε, επί τη βάση της μελέτης, ότι η σύμβαση της Χάγης του 80 έπεσε θύμα της επιτυχίας της. Ο μηχανισμός της αυτόματης επιστροφής ήταν τόσο αποτελεσματικός που ενίσχυε ε, την χρήση του και σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλεπόταν να ισχύζει. Βλέπουμε ότι πρώτα-πρώτα η κλασική περίπτωση ήταν το να καλυφθεί η περίπτωση της απαγωγής του ανηλίκου από τον ε, πατέρα που ήθελε οριστικά να αποσπάσει αυτό το, το ανήλικο από την μητέρα του. Υπήρξε ε, πρόθεση σύναψης διμερών συνθήκων μεταξύ κρατών μελών αλλά και με τρίτες χώρες και κυρίως ε, και με αραβικές χώρες με την Γαλλία. Λίβανο, Αίγυπτο, Μαρόκο γιατί εκεί είναι όλος διάφορη η θέση της γυναίκας σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο των χωρών εκείνων. Οπότε και τώρα είχαμε τελικά μία ερμηνεία εξελικτική της ρύθμισης. Ούτως ώστε τελικά η πλάστιγκα έγινε υπέρ του γονέα ο οποίος είχε την γονική μέρημνα και επιμέλεια του ανηλίκου. Και έτσι τώρα καλύφθηκε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής κατοικίας του ανηλίκου σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνήσει και ο άλλος γονέας. Επομένως τώρα άλλαξε και η σύλληψη του δικαστή η αντίληψη του δικαστή τώρα θα έπρεπε να λάβει υπόψη και τις λιγότερο άμεσες ανάγκες επιστροφές του ανηλίκου και έτσι τώρα δημιουργήθηκε όλο αυτό το θλιβερό βουνό νομολογίας το οποίο εμφανίστηκε ε, προς εκδίκαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των δικαιωμάτων. Πάντως, ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α που ενισχύει το μηχανισμό της άμεσης επιστροφής είναι ένα βήμα πρόοδου. Βλέπετε τώρα εδώ ποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε. Έχουμε τώρα το, την ε, παραβίαση των δικαιωμάτων της επίσκεψη από τον ένα γονέα. Είδαμε ότι ε, είχαμε περιπτώσεις τέτοιες στην Ιρλανδία, ε, είχαμε παγωγή από έναν θείο, ε, που πήγε τον ανήλικο στην Αίγυπτο στον πατέρα. Επίσης ε, έχουμε τώρα την, ε, την περίπτωση του γονέα που έχει επιμέλεια και γονική μέρημνα και, και που εμποδίζει την συμμετοχή του άλλου γονέα στην ανατροφή του παιδιού. Και είδαμε εδώ πέρα στην Λιθουανία ότι είχαμε παραβίαση του άρθρου 8 ε, του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, κατά τρίτον, έχουμε όλες τις περιπτώσεις απαγωγής που γίνονται προς συμφέρον του ανηλίκου ε, και πολλές φορές ε, έχουμε κάποιο είδους απαγωγής για λόγους άμυνας. Είναι οι εξαιρέσεις της ε, σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 13. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται άμεση αντίδραση. Πρόκειται για περιπτώσεις που συμβαίνουν συνεχώς. Πρόκειται για όλα αυτά που έχουν καταγραφεί στις στατιστικές. και σε αυτή την περίπτωση είπαμε ότι υπάρχει αύξηση των περιστατικών. Πρόκειται επομένω για κατά κάποιο τρόπο τη συνέπεια της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Είναι λοιπόν το δικαίωμα της ε, επίσκεψης οπότε παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Ή επίσης ο γονέας ο οποίος έχει την γονική μέρημνα και επιμέλεια καταχράται του δικαιώματός του, παίρνει το παιδί και πάει σε άλλη χώρα. Θεωρείται ότι αυτή η μετακίνηση των ελίκου είναι παράνομη. Επομένως έτσι διαρριγνεί αυτός ο γονέας την σχέση το παιδιού με τον άλλο γονέα. Ο μηχανισμός τώρα της άμεσης επιστροφής είναι τώρα τόσο πολύπλοκος σε αυτές τις περιπτώσεις που οι δικαστές διστάζουν να διατάξουν την ε, επιστροφή. Έχουμε τις εξαιρέσεις της σύμβασης της Χάγης πάντοτε μπορεί κανείς να σταθμίσει ποια είναι τα υπέρτερα συμφέροντα του ανηλίκου και σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να γίνει στάθμιση επομένως του ποιο είναι το υπέρτερο συμφέρον του ανηλίκου. Και πάντα υπάρχει τώρα αυτή η ανισορροπία. Ότι ποιος γονέας βρίσκεται συμπατριώτης με τον δικαστή που κρίνει την περίπτωση και ο άλλος πολλές φορές είναι μετανάστης στη χώρα εκείνη που δικάζεται η περίπτωση και είναι το θέμα της ε, μη άρτιας γνώσης του δικαίου ή της γλώσσης ή της ε, κοινωνικής ένταξης του ενός από τους δύο γονείς. Αυτό πολλές φορές επηρεάζει επομένως την κρίση του δικαστή. Πρόκειται ουσιαστικά για σύγκρουση δύο νόμων τάξεων. Τώρα, για να αποφύγουμε τέτοιες συνέπειες θα πρέπει να βρεθεί ε, μια λύση, ένα σύστημα που να βασίζεται σε κάποια διάκριση των περιπτώσεων πιο ε, ακραίων και εκείνων που απλώς χρειάζονται κάποια στάθμιση. Άρα χρειάζεται να υπάρξει κάποιο φιλτράρισμα. Ανάλογα με το πόσο ακραία είναι η περίπτωση της απαγωγής. Επομένως, στις ακραίες περιπτώσεις χρειάζεται αποτελεσματικότητα και μεγάλη ταχύτητα αντίδρασης. Πάντα τσαθμίζονται λοιπόν τα συμφέροντα του ανηλίκου και είναι δεδομένο να ληφθούν κάποια ε, ασφαλιστικά μέτρα προστασίας του ανηλίκου. Τώρα, οι περιπτώσεις όμως που δεν εντάσσονται ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να κριθούν διαφορετικά από τους δικαστές γιατί ο δικαστής της συνήθους κατοικίας θα πρέπει να καταλήξει σύμφωνα με το άρθρο 15 της ε, Σύμβασης των Βρυξελών. Θα πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία ουσιαστικά μεταξύ των δικαστών των δύο χωρών των δύο γονέων. Όμως, λέγεται ότι χρειάζεται κάποιος υπέρεθνικος δικαστής. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να λάβει αυτό τον ρόλο. Θεωρούμε ότι αυτή η μελέτη βοηθά την προβληματική σε ένα θέμα τόσο περιπλόκο και τόσο λεπτό. Σας ευχαριστούμε για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Και τώρα δώσουμε απευθείας τον λόγο στον κύριο Λιβαδόπουλο που είναι δικηγόρος και διαμεσολαβητής σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα να περάσω στην παρουσίασή μου. Θα ήθελα να μιλήσω για την διαμεσολάβηση σε διεθνείς υποθέσεις απαγωγής παιδιών. Δούμε ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η διαμεσολάβηση, ε, Βρυξέλλες 2α ε, πρώτα απ' όλα ε, και η σήμαση της Χαγής του 1980 προβλέπουν διαμεσολάβηση σε τέτοιες υποθέσεις και συνεργασία των κεντρικών αρχών προς μια, έναν εξοδικαστικό φιλικό διακανονισμό σε διασυνοριακές υποθέσεις απαγωγής παιδιών υπάρχει και η Οδηγία 52 του 2008, βάσει της οποίας μπορούν να αποφασίσουν οι δικαστές να καλέσουν τους γονείς ε, να προσφύγουν και να καταλήξουν σε έναν διακανονισμό και ε, θα μπορούσε ενδεχομένως να επιληθεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Υπόθεσης. Πώς λειτουργεί αυτή η διαμεσολάβηση. Λοιπόν, στις διασυνοριακές ε, υποθέσεις, ε, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η διαμεσολάβηση, ε, κατά τη διάρκεια ή πρώτης διαφοράς, οι περισσότερες υποθέσεις που φτάνουν στο δίκτυό μας είναι πριν από την ακρόαση στο δικαστήριο, στο δικαστήριο που αποφασίζεται η πρώτη διαφορας οι περισσοτερες υποθεσεις που φτανουν στο δικτυο ή όχι του παιδιού σε αυτό το στάδιο λοιπόν και η διαμεσολάβηση γίνεται σε ουδέτερο μέρος και φυσικά στο κράτος όπου κρατείται ε, το παιδί ή τα παιδιά ε, προσωρινά. Φυσικά τα μέρη και οι διαμεσολαβητές και όχι οι διαμεσολαβητής στο πληθυντικό διότι χρησιμοποιούμε το εξή μοντέλο που βασίζεται στην έννοια της συνδιαμεσολάβησης. Θα το εξηγήσω σε λιγάκι η επικουρούνται από τους δικηγόρους των μερών, αλλά μέσω τηλεφωνικής γραμμής Skype, email επικοινωνούν, δεν είναι παρόντες όταν μιλούμε για την ε, Συμφωνία για τη Διαμεσολάβηση. Υπάρχουν λοιπόν οι διαμεσολαβητές επιτόπου και ε, τα μέρη σε κοινέ ε, μικτές και χωριστές ακροάσεις. Ε, περισσότερες είναι οι μικτές κατά τη διάρκεια της και ο στόχος είναι να βρεθεί μια συνενετική λύση από τους διαδίκους. Φυσικά γίνεται αυτό σε εθελούσια βάση και τηρείται χεμήθεια. Πριν τη διαμεσολάβηση, τι πρέπει να κάνει ο διαμεσολαβητής, ε, να εξετάσει, να ε, κάνει τις εξακριβώσεις για την υπόθεση, ώστε να αποφασίσει αν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαμεσολάβησης. Ε, και με το που γίνεται αυτό, στη συνέχεια προβαίνουν στις απαιτούμενες επαφές για να αποφασίσουν πού πρέπει να λάβει χώρα και με ποιο τρόπο που να λάβει η χώρα η διαμεσολάβηση, αυτό σε συμφωνία με τους διαδίκους και τους συνηγόρους τους. Αυτή είναι η πρώτη φάση της διαμεσολάβησης, γίνεται η παρουσίαση, η συμφωνία, η συνένεση, η διαμεσολάβηση. Μετά αποστέλλεται η ημερήσια διάταξη, τα θέματα που θα εξεταστούν, στη συνέχεια διερευνούνται οι ανάγκες, οι επιθυμίες των διαδίκων η έρευνα της υπόθεσης, μετά εξετάζονται οι λύσεις για την, οι πιθανές λύσεις σε περίπτωση απαγωγής παιδιού θα πρέπει να αποφασιστεί και ο τόπος διαμονής ε, αν θα παραμείνει επί τόπου το παιδί ή θα πρέπει να επιστρέψει στην χώρα ε, από την οποία απήχθηκε. Το πέμπτο στάδιο είναι το τελευταίο στάδιο όπου λαμβάνεται η απόφαση αυτή η συνειδητική απόφαση. Υπάρχουν πολιτισμικές ε, διαφορές ε, που απειλούν ε, αυτές τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, αυτές οι διαφορές ενδεχομένως να μην φαίνονταν να ήταν τόσο αισθητέ όσο έβαινε αισίως η σχέση, αλλά όταν επιδεινώνεται η σχέση εμφανίζονται πιο έντονα. Θα τις περισσότερες φορές ε, θέλει κάποιος να γυρίσει στην χώρα πρέλευσης του μετά το χωρισμό και θέλει να τον ακολουθήσει το παιδί και τότε συμβαίνει η απαγωγή και ο γονέας που μένει πίσω ε, νιώθει αβοήθητος, ε, νιώθει οργισμένος, και φυσικά σε περίπτωση, στην περίπτωση απαγωγής φοβούνται την απώλεια του παιδιού και οι δύο γονείς και το παιδί μένει δέσμιο ανάμεσα στους δύο, παγιδευμένο ανάμεσα στους δύο. Ε, αλλά για να περάσουμε στα συγκεκριμένα ζητήματα, το βασικότερο ζήτημα και με το οποίο ξεκινούμε τη διαμεσολάβηση είναι να αποφασίσουμε αν θα επιστρέψει ή δεν θα επιστρέψει το παιδί. Μόλις βρεθεί μια λύση από τους γονείς τότε ε, προχωρούν και μιλούν για το μελλοντικό τόπο διαμονής, ε, για ε, το δικαίωμα επίσκεψης, ε, για τη γονική επιμέλεια, μέρημνα, το, το πότε, πού θα περνάει τις διακοπές, το παιδί, ποιος θα πληρώνει τις διακοπές, ποιος θα βγάζει τα αεροπαρικά εισιτήρια, σε, σε σχέση με την δίγλωση, η διαπαιδαγώγηση, η ανατροφή του παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί ή τα παιδιά είναι σημαντικό για τους δύο γονείς να ανατρέφονται βάσει του συστήματος της χώρας τους και ορισμένες φορές όταν ε, ε, διευθυντούνται αυτά τα ζητήματα, περνάμε στο χωρισμό, στο διαζύγιο, στο διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων. Αν δηλαδή δεν έχουν ήδη πάρει διαζύγιο, μπορούν ήδη να αρχίσουν να συζητάνε και αυτά τα ζητήματα. Φυσικά το πιο σημαντικό για τους γονείς, ε, όπως είπα, είναι ε, αν θα επιστρέψει ή όχι το παιδί στην χώρα από την οποία απήχθη. Το πλαίσιο τώρα, ε, μέσα στο οποίο μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία διαμεσολάβησης, η κεντρική αρχή, ο δικαστής, οι διαμεσολαβητές, οι συνήγοροι, οι διάδικοι μπορούν να ανακοινήσουν την διαδικασία. Υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα Σα είπα κυρίως πρώτης ακροματική διαδικασίας στο δικαστήριο, τότε αποφασίζουν ε, κατά κανόνα τα ζευγάρια να προσφύγουν σε τέτοια διαμεσολάβηση. Ε, είναι πολύ χρονοβόρα η προετοιμασία, πρέπει να γίνουν τα ταξίδια, να μιλάνε με τους συνηγόρους τους, χρειάζονται δύο-τρεις ημέρες για τις ε, μεικτές ακροάσεις, ε, υπάρχει κλιμάκωση της έντασης, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, νιώθουν πικρία, θυμό, ε, φοβούνται να μην χάσουν το παιδί, ε, ε, αβεβαιότητα σε σχέση με την έκβαση της διαδικασίας. Τι, ποιο μοντέλο χρησιμοποιούμε τώρα για τη διαμεσολάβηση. The model we use to do the mediation is, a. Uh, το μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι η σύνδια μεσολάβηση, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Τι σημαίνει αυτό οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να προέρχονται από τους δύο πολιτισμούς, αν θέλετε. Δηλαδή, ε, από τις δύο χώρες από τις οποίες ε, προέρχονται και οι διάδικοι. Άμα είναι ε, από την Ελλάδα και τη Γερμανία θα έχουμε δύο διαμεσολαβητές αντίστοιχα από την Ελλάδα και τη Γερμανία και οι δύο γλώσσες και τα δύο φύλλα επίσης εκπροσωπούνται για να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση ε, διαφορετικό επίσης ε, οικονομικό, νομικό, επαγγελματικό υπόβαθρο. Φροντίζουμε ε, πάντοτε βεβαίως να, να ε, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του παιδιού. Για να δείτε στην πράξη πώς είναι μια τέτοια διαμεσολάβηση. Στα δεξιά σα βλέπετε τους δύο διαμεσολάβητέ και στο αριστερό σα χέρι είναι το ζευγάρι και στη μέση είναι ε, ο διερμηνέας ή η διερμηνέας. Η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Αν θέλει το ένα μέρος να μιλήσει τη γλώσσα του ή και μία τρίτη γλώσσα μπορεί να ζητήσει της υπηρεσίας ενός ε, ε, διερμηνέα. Ε, το 2012 συγκροτήθηκε το δίκτυό μας, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η ΜΚΑ Μικρονίκ από τη Γερμανία, το Child Focus από το Βέλγιο, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν και το Ολλανδικό Κέντρο για τις Διασυνοριακές Απαγωγές των Παιδιών είναι τα συμβαλλόμενα μέρη του δικτύου. Έχουμε περίπου 70 διασωμελαβητές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώτη φορά κάναμε ε, ένα ενοποιημένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων δημιουργήθηκε στο δίκτυο. Μας παρέπεμψαν ε, σταδιακά όλα είναι και περισσότερες υποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, όπως συμβαίνει συνήθως, ε, ένα mail στους ε, στέλνουμε ένα mail σε όλους τους διαμεσολαβητές, ανεξαρτήτως χώρας, άμα είναι ένας Ιταλός υπήκος, παραδείγματο χάρη, ε, γίνεται η επαφή με τον ε, Ιταλό διαμεσολαβητή και αν το άλλο μέρος είναι από τη Λιθουανία, παραδείγματο χάρη, ο Ιταλός διαμεσολαβητής θα ε, τηλεφωνήσει, ε, θα έρθει επαφή με τον συνάδελφο ή τη συνάδελφο από τη Λιθουανία για να προσπαθήσει να ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες για τη διαμεσολάβηση. Ε, το Meet the Child Fox και το Missing ε, Child Europe ε, συνεργάζονται λοιπόν στο δίκτυο αυτό. Το Missing Child Europe είναι στις Βρυξέλλες. 50 ώρες εκπαίδευση έχουμε δυσίως για τους νέους διαμεσολαβητές και εντατικά μαθήματα για τα μέλη μας. Το ε, the Voice of the Child in Mediation, αυτό είναι το μελλοντικό μας πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών υποθέσεων και για τη διαμεσολάβηση και φυσικά η ψυχολογική διάσταση, δηλαδή η προστασία των, ε, του ευζήν και των συμφερόντων του παιδιού. Μπορείτε στο site μας να βρείτε τις ε, περισσότερες πληροφορίες αν το επιθυμείτε. Σας ευχαριστούμε κύριε Λιβαδόπουλο. Τώρα... Ο κ. Χάνς Φουνλούν από το Ινστιτούτο Διεθνού Δικαίου και με αντιπρόεδρο τη ε, πρώην Σύμβαση τη Χάγη για το Διεθνέ Ιδιωτικό Δίκαιο και ο Μέση Ισότο, προστάμενο μονάδα πολιτική δικαιοσύνη, γραμματέα δικαιοσύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μεγάλη τιμή είναι εμφανίζομαι σε αυτή την ε, Επιτροπή για το Κοινοβούλιο και εγώ αναφέρομαι στις Βρυξέλλες 2, αλλά μόνο σε θέματα αγωνικής ευθύνης. Ο αρχικός κανονισμός Βρυξέλλες 2 πραγματεύτηκε τα θέματα αυτά μόνο σε ό,τι αφορά το πλαίσιο του διαζυγίου. Αλλά υπήρξε μία αντίληψη από πλευράς κάποιων κρατών μελών ότι οι διατάξει ε, τη συνθήκη για την απαγωγή των παιδιών δεν ε, είχαν ληφθεί υπόψη στο κεφάλαιο 2 στη σελίδα 831 του δευτέρου εγγράφου. Σημεία 2 και 3 πραγματεύεται ακριβώς αυτή την αντίληψη. Είναι σημαντικό να τονίσουμε εξ αρχής λοιπόν ότι η γονική ευθύνη και οι απαγωγές παιδιών δεν αποτελούν ε, φυσικά αποκλειστικά ευρωπαϊκό φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο θέμα. Υπάρχει λοιπόν ένα παγκόσμιο πλαίσιο το οποίο αποτελείται από τη σχετική συνθήκη του ΟΗΕ, τη συνθήκη της Χάγης και τη ε, συνθήκη του 86 για την προστασία των παιδιών. Τα κράτη-μέλη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν, ε, είχαν προσπογράψει την ε, συνθήκη του 86 εδώ και καιρό. Και η συνθήκη του 96 ισχύει για όλες ε, τις χώρες εκτός από την Ιταλία. Αλλά η σύνοδος ε, της ε, Ρώμης την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισε να προσυπογράψει την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν. Αυτό θα αυξήσει λοιπόν την αποδοχή του διεθνούς πλήσεου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη του 96, όπως η Ρωσία, το Μαρόκο, η Δανία, και Επίσης, η συνθήκη του 96 παρέχει του ρόλου για το... παρέχει τις ε, διδάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Είναι λοιπόν ε, καλή στιγμή να ξανακοιτάξουμε τι προβλέπουν οι Βρυξέλλες 2 υπό το πρίσμα αυτού του διεθνούς ε, πλαισίου. Η συνθήκη του 96 ήταν ουσιαστικά η πηγή έμπνευση για τις Βρυξέλλες 2, αλλά οι Βρυξέλλες 2 έχει διάφορα σημαντικά επιπλέον στοιχεία σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ιδιαίτερα επιστροφής. Όχι μόνο ενισχύει τις ε, αρμοδιότητες του δικαστηρίου ε, προέλευσης που γίνεται και η συνθήκη του 96, αλλά μειώνει και τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου του τόπου προορισμού. Αυτό είναι προβληματικό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και αυτό αναφέρεται και στην ελβετική μελέτη και αυτό τονίζει πόσο σημαντική είναι η ισορροπία μεταξύ των αξουσιών των δύο δικαστηρίων. Στο κεφάλαιο 2 θα βρείτε τις εξελίξεις αυτές. Η κλασική περίπτωση είναι αυτοί που είχαν κατά νου που είχαν η συνθήκη του 96 και Βρυξέλλες, δύο ήταν του γονέα που δεν έχει την κυδαιμονία. Τα πράγματα λοιπόν έχουν περιπλοκεί και σε δύο-τρία στα δύο-τρία των περιπτώσεων ο γονέας που κάνει την απαγωγή είναι ο γονέας ο οποίος φροντίζει το παιδί. Είτε η μητέρα η οποία κατηγορεί για βία ενδοοικογενειακή. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε πιο πολύ προσοχή από ό,τι στο παρελθόν στον κίνδυνο που ενέχεται για το παιδί, για την ασφάλεια του παιδιού. Επίσης δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο την άποψη του παιδιού για την επιστροφή και τώρα βλέπουμε ότι ο γονέας που έχει μείνει πίσω πιο συχνά από το παρελθόν εξαρτάται από τη συνθήκη και από τον κανονισμό. Όχι τόσο για να έχει την επιστροφή του παιδιού μόνιμα, αλλά για να ισχύσουν τα δικαιώματα πρόσβασης του. Όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει σε μία μετατόπιση, αν θέλετε, και αυτή η μετατόπιση έχει οδηγήσει σε επίκριση της συνθήκης και στο κεφάλαιο λοιπόν αυτό, στο κεφάλαιο 2, εξετάζονται αυτό. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί ότι όταν τίθεται θέμα επιστροφής θα πρέπει να ακούμε τα επιχειρήματα με προσοχή και οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένες, να υπάρχουν αποδείξεις προστασίας του παιδιού αν, αν υπάρχει και έχετε κίνδυνος και η επιστροφή δεν θα πρέπει να είναι αυτόματη. Επίσης, και η συνθήκη έχει ασχοληθεί, το συνέδριο έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια κοινή άποψη ότι χρειάζονται και συνοδευτικά μέτρα. Η επικύρωση της συνθήκης της 96 λοιπόν για μεγαλύτερη προστασία του παιδιού. Δημιουργήθηκε μια ομάδα για να οδηγήσει καθοδήγηση στα δικαστήρια για την ερμηνεία της συνθήκης και δημοσιεύτηκε και ένα κατάλογο για τη διαμεσολάβηση μεταφρασμένου σε όλε τι γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. χάρη στην υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πολύ ευγενική υποστήριξη. Ποια ήταν λοιπόν η αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτέ τι νέε εξελίξει. Αφενό έχει υποστηριχθεί ασφαλώ η νέα πρωτοβουλία. Από την άλλη, μα προκαλεί εντύπωση ότι έχει γίνει πάρα πολύ λίγη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι αλλαγέ αυτέ. Το δικαστήριο έχει αναφερθεί στο, στη συνθήκη και στο μηχανισμό επιστροφή ως αντικίνητρο και ως ε, κίνητρο να κάτσουν να μιλήσουν οι δύο γονείς, αλλά δεν έχει αποφανθεί, από όσο ξέρω, το δικαστήριο γιατί υπάρχει πρόθεσμο αντίκτυπο της επιστροφής στο κεφάλαιο 3 από τη σελίδα 20 και εξή μας ε, προσπαθεί να δώσει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για τον κανονισμό για να εναρμονιστεί πιο πολύ στο παγκόσμιο προσκήνιο, ιδιαίτερα στη συνθήκη του 96, αλλά να προσαρμοστεί και στη μετατόπιση τη νοοτροπία. Βλέπετε, στη σελίδα 39-33 έχουμε ε, το... το παράρτημα. Και σημαντικό λοιπόν είναι να λεφτούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, αυτή μετατόπιση και η αλλαγή τη νοοτροπία. Οι προτάσεις ε, δεν έχουν ως σκόπο να ξαναγράψουν τον κανονισμό. Σεβόμαστε τι αρχές του κανονισμού. Υπάρχουν δύο κατηγορίε ε, προτάσεων. Αφενό, οι προτάσεις εκείνε που σκοπό έχουν να εναρμονιστεί πιο πολύ ο κανονισμό στο πλαίσιο και να προσαρμοστεί στην αλλαγή αυτή των εξελίξεων και κατά δεύτερον υπάρχουν πολύ καλοί κανόνε στον ίδιο τον κανονισμό που υπερβαίνουν το ίδιο το πλαίσιο και που θα μπορούσαν επιπλέον να τονιστούν. Να ξεκινήσουμε την πρώτη ομάδα. Προτάσει λοιπόν γιατί να ενερμονιστεί ο κανονισμό στην συνθήκη του 96. Έχουμε στην κεφάλαιο 8 την πρόταση και πιο σημαντικά έχουμε και την πρόταση τροποποίησης του κεφαλαίου του άρθρου 10 να εισαχθεί νέος ε, ορισμός για τα προστατευτικά μέτρα. Γιατί στις Βρυξέλλες 2 ε, οι νομοθέτες εμπνεύστηκαν από το Βρυξέλλες 1, που ήταν πιο πολύ για εμπορικά ζητήματα. Αλλά αυτό διαφέρει από τα οικογενειακά ζητήματα. Και έχουμε λοιπόν τρία προβλήματα σε ό,τι αφορά το άρθρο 20. Δεν υπάρχει ενιαία βάση δικαιοδοσία. Το δικαστήριο που αποφασίζει την επιστροφή μπορεί να επιβάλλει προστατευτικά μέτρα που θεωρεί το ίδιο σωστά. Κατά δεύτερον, τα μέτρα αυτά, αν υπάρχουν, μπορούν να ληφθούν κατά του παιδιού στην δικαιοδοσία του δικαστηρίου και όχι στη δικαιοδοσία άλλων. Και τρίτον, τα προστατευτικά μέτρα αυτά πρέπει να αναγνωριστούν στο δικαστηρίο προέλευσης. Άρα, αν κάποιος εξετάσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει ένα παιδί, αλλά το συνδέσει αυτό μόνο με προστατευτικά μέτρα κατά ενός πατέρα, για παράδειγμα, που ε, ακόμα τα χειρίζεται το παιδί του, δεν μπορεί να επιβάλλει τα μέτρα αυτά στην άλλη χώρα. Άρθρο 11, 6 και 8 και 42 βασίζονται στην ιδέα ότι οποιαδήποτε άρνηση επιστροφή ε, του παιδιού του δικαστηρίου δίωξη μπορεί να ε, αναιρεθεί από το δικαστήριο προέλευση. Γιατί ουσιαστικά εδώ Υπάρχει το αντίστροφο αυτό που αυτό συμβαίνει συνήθω. Μία απόφαση του δικαστηρίου δίωξη μπορεί να ανατραπεί από το δικαστήριο τη προέλευση, τη χώρα προέλευση. Αυτό ενδεχομένω να μην είναι και το πιο φυσιολογικό, γιατί αποθαρρύνει ασφαλώ και δεν δίνει κίνητρα στο δικαστήριο όπου γίνεται η δίωξη. Το δικαστήριο δίωξη θα είναι αυτό που καλείται να αποφασίσει για το, τα συμφέροντα του παιδιού. Και το δικαστήριο της χώρας προέλευσης να αποφασίσει για θέματα δαιμονία. Είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά. Να μην συγχέονται. Το δικαστήριο λοιπόν δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα πολύ φοβάμαι, γιατί αποφάνθηκε ότι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου της χώρας προέλευσης μπορεί να ληφθεί επίσης σε διάφορες περιστάσεις, σε διάφορες φάσεις. Άρα μπορεί να διαταχθεί η επιστροφή του παιδιού και τελικά να έρθει μια τελική απόφαση ότι θα πρέπει ξανά να φύγει το παιδί. Και να πάει στο, στη χώρα όπου, ήταν, ε, όπου είχε μεταφερθεί κατά την απαγωγή του. Διαγραφή του άρθρου 42 ενδεχομένω. Δεν ξέρω να συνεχίσω ή θέλετε να σταματήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ το άρθρο 42. Εξαρτάται, λέει η πρόεδρο. Εξαρτάται από το γείτονά σα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είμαι σύντομο, θα είμαι σύντομο. Άρα, ω εκ τούτου, υπάρχει πρόβλημα και στο άθρο 42. Γιατί προβλέπει την εφαρμογή της ε, επιστροφής που έχει αποφασίσει το δικαστήριο και κανένας λόγος άρνησης ούτε καν το συμφέρον του παιδιού δεν ισχύουν εδώ. Και αυτό πραγματικά υπερβαίνει τα όρια. Δεν είναι και απαραίτητο άλλωστε, γιατί οι διατάξει του 1, 2, 3 του ίδιου κεφαλαίου, του ίδιου άρθρου, αποτελούν ένα πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω αυτό το επιχείρημα, αυτό το πείραμα. Και για το 44 το άρθρο θα μπορούσαμε να έχουμε αμφιβολίες. Ε, όπου έχουμε την πρόβλεψη επιστροφής του παιδιού χωρίς να υπάρχουν απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την ασφάλεια του παιδιού. Προτάσεις τώρα. Πού, μπορεί, πού πρέπει να πάμε λίγο παραπάνω από αυτά που προτείνει ο κανονισμός. Πρόταση για ε, επανατοποθέτηση μετά από σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 12 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Πρόταση να ενισχυθεί να διευρυνθούν οι διατάξει που αναγκάζουν το δικαστήριο να αποφασίσει σε έξι μήνες. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν χρονικό περιθώριο. Και τέλος μια διάταξη που προτείνει η διαμεσολάβηση να ενταχθεί στο πλαίσιο του κανονισμού όπως γίνεται ήδη σε κάποιες χώρες όπου τα δικαστήρια ε, πριν ε, αποφανθούν ε, εξετάζουν το ενδεχόμενο διαμεσολάβηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ευχαριστώ που μου δώσατε και λίγο παραπάνω χρόνο να μιλήσω. Thank you very much. Um, I speak from the Commission's perspective. Ευχαριστώ πολύ. Να σα πω από πλευρά τη ε, Γενική Διεύθυνσης για θέματα Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την ε, εφαρμογή του κανονισμού Βρυξελών 2α, το επίκεντρο των προβληματισμών ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τα όσα είπαμε τώρα, δηλαδή, τα όσα λέμε τώρα, πολύ χρήσιμο για μα και όπω πάρα πολύ εξημό θα γνωρίζετε ότι στον κανονισμό 2α τώρα έχουμε μία ισχύ του για μία δεκαετία και τα τελευταία χρόνια είχαμε κάποιε διαφορέ κοινωνικού δικαίου, οι οποίε αυξήθηκαν, είδαμε τα στατιστικά, μα τα παρουσίασαν πριν από λίγο και, και γνωρίζουμε πόσο δύσκολο κανεί είναι να αποσπάσει τέτοια στατιστικά στοιχεία ε, τα έχουν παρακολουθήσει από κοντά, αλλά αυτό το οποίο είναι σίγουρο μέσα σε έναν ολοένα και πιο μεταβαλλόμενο κόσμο ότι όλα αυτά τα φαινόμενα αυξάνονται και έχουμε 15 εκατομμύρια πολιτών οι οποίοι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα που δεν είναι η χώρα προελευθής οπότε κάθε χρόνο έχουν περίπου 140.000 ε, διεθνή διασυνοριακά διαζύγια αυτό σημαίνει ότι αυτές οι διασυνορια, οι οικογένειες που περνάνε τα σύνορα ε, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή τη προβληματική σήμερα. Οπότε βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σωστικό το πρόβλημα για τόσο, τόσο κόσμο. Οπότε ε, ε πάρα πολύ σωστά συζητούμε τώρα το θέμα αυτό και βλέπετε ότι οι πολιτικέ ε, καθημερινέ γραμμέ παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο Γιούγκερ πέρσι και είδατε τι γίνεται όσον αφορά τη δικαιοσύνη για δημιουργία δικαιώματα, κάτι το οποίο βασίζεται στην αμοιβή εμπιστοσύνη και πρόκειται για μία από τι 10 βασικέ πρωτεύουσε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω πολίτε που κινούμε στο εξωτερικό και παντρευόμαστε και αποκλούμε παιδιά, βλέπουμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η δικαστική συνεργασία και βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση επί τη βάση ε, της εμπιστοσύνης ε, φτιάχνοντας αυτές τις ε, γέφυρες μεταξύ των ε, νόμων τάξεων ούτω ώστε να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε την αμοιβαία, τον, την αμοιβαία εμπιστοσύνη αλλά βέβαια αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει είναι να προσπαθήσουμε να ακούμε τη φωνή όλων και να, έτσι να πλουτίζουμε την ευθοσύνη μας. Ο κανονισμός των Βρυξελών ακριβώς ε, έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτή την δικαστική συνεργασία και είναι πάρα πολύ στο το Κοινοβούλιο και Κομισιόν προσέχουν πάρα πολύ το πώς ε, προχωρούν τα πράγματα και αυτό εξηγεί γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη μέση μιας διαδρομής ούτως ώστε να αναθεωρήσει ε, την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. για την πρώτη αναθεώρηση. Και μια που έχουμε εδώ όλους αυτούς τους εμπειρογνώμονες, όλους όσους βρίσκονται εδώ, θα πρέπει και εμείς να τους σας πούμε ποια είναι τα πρώτα μας συμπεράσματα και να ακούσουμε και από εσά ε, τις ιδέες σας, τις ε, θέσεις σας. Οπότε, χωρίς καθυστέρηση να σας αναφέρω το ότι τον Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε μια έκθεση και κατέληξε στο ότι ο κανονισμός ωφέλησε ουσιαστικά τους Ευρωπαίους ούτω ώστε να ρυθμιστούν καλύτερα αυτές οι ένδικες διαφορές που αφορούν τα ζητήματα αυτά οικογενειακού δικαίου. Συνεργασία εθνικών αρχών να αποφύγουμε παράλληλες δίκες και παράλληλες δικαστικές αποφάσεις. Πολύ σημαντικέ βέβαια διατάξει για την επιστροφή των παιδιών. Σημαντική λειτουργία τη αποτροπή. Να προσέξουμε τα στατικά στοιχεία. Φυσικά και διάβασα προσεκτικά το κείμενο του κ. Φανλόν. Πάντω. όταν θεσπίστηκε αυτός ο κανονισμός, υπήρξε ακριβώς αυτή η πρόθεση του νομοθετή. Να δούμε κατά πόσον η αποτροπή λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Έχουμε όλα τα πλέον επομένω του κανονισμού των Βρυξελών, αλλά από την άλλη μεριά διαπιστώθηκαν και από την έκθεση κάποια μειονεκτήματα. Ιδίω όσον αφορά τα θέματα δικαιοδοσία, τι γαμικέ διαφορέ, αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Επίση, η κατάργηση του εξεκουάτορ, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα πλαίσια των συμφερόντων του παιδιού, που πολλές φορές η χρονική πίεση είναι μεγάλη. Επίσης ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί η συνεργασία των εθνικών αρχών. Και αυτή η συνεργασία είναι η καρδιά της ρύθμισης και στον κανονισμό του Βρυξέλλες 2. Πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής του νόμου. Οπότε και σύμφωνα με την έκθεση δεν πάνε τα πράγματα τόσο καλά, δεν υπάρχει τόσο εύρυθμη λειτουργία του συστήματος όπως θα περιμέναμε. Επομένως, είπαμε ότι το καλύτερο είναι το να γίνει μια διαβούλευση. Η διαβούλευση έγινε, ολοκληρώθηκε το θέρος του 2014, είχαμε μεγάλη συμμετοχή από νομικούς, δικηγόρους, δικαστικούς, ε, απλούς πολίτες, διαπιστώθηκε το πώς βλέπουν την λειτουργία της ρύθμισης. Βεβαίως ήταν ε, ανάμεικτα τα αισθήματα του κόσμου, θετικά και αρνητικά. Θεωρήθηκε ότι για τέτοιες διασυνοριακές γαμικές ε, οικογενειακές διαφορές βοηθά αυτός ο οργανισμός. Εάν επομένω εφαρμοστεί ο κανονισμό με το πνεύμα με το οποίο θεσπίστηκε ότι, ότι βοηθά. Όμως, από την άλλη μεριά, βγήκαν και κάποια προβλήματα. Δεν υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού από όλα τα κρατημέλη και αυτό πολλές φορές οφείλεται στο ότι δεν είναι σαφής ο ίδιος ο κανονισμός. Ας πούμε σε περιπτώσεις απαγωγών πάρα πολλοί ετώνησαν ότι υπάρχει δυσκολία λήψης απόφασης μέσα στην προθεσμία των έξι εβδομάδων που προβλέπεται. Κάποιοι δικαστές είπαν ότι δεν είναι τόσο εύκολη η εκπαιρέωση των αιτήσεων επιστροφής. Πολλές φορές είπαν ότι είναι μεγάλη ποικιλία των διαφορετικών δικαστηρίων στα οποία υποβάλλονται αυτές οι αιτήσει επιστροφής των ενηλίκων. Άρα θα έπρεπε να βρεθεί ένα δικαστήριο, να εξειδικευθεί κάποιο δικαστήριο. Διαπιστώθηκε ότι αυτό θα διευκόλυνε. Και αυτό θα βοηθούσε να ληφθεί απόφαση μέσα στις 6 εβδομάδες. Επίσης, όσον αφορά την απόφαση επιστροφής, θα έπρεπε να είναι η ρύθμιση πιο ξεκάθαρη. Τα είπε ο κ. Φανλόν. Η εφαρμογή του κανονισμού γίνεται με κάποιε διαδικασίε κοινοτενή που δεν ωφελούν. ακριβώ για τι περιπτώσει αυτέ έχει σημασία ο παραγόν χρόνο. Να, που θεωρούμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μας. δεν είναι δυνατόν με έναν κανονισμό να λύνονται όλες ατομικά οι αλλά μπορούμε να δούμε αντίστροφα από την κάθε περίπτωση, από τα προβλήματα που ανακύπτουν, που επιδέχεται βελτίωση ο κανονισμός. Δεν μιλούμε για επανάσταση στην νομοθεσία απλώς, λίγο-λίγο να βελτιώνουμε αυτό το οποίο ήδη έχουμε φτιάξει. Να σας πω σε ποιους τομείς θεωρούμε ότι πρέπει κάτι να γίνει. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τις γαμικές διαφορές. να μπορούν οι σύζυγοι να διαλέξουν το δικαστήριο όπου θα εκδικαστεί το διαζύγιο, όπου θα συζητηθεί το διαζύγιο. Άρα να τους ενθαρρύνουμε να συνεργαστούν, να βρουν κάποια συμβαστική διαφορά. Αυτό γίνεται και σε άλλες συγκρίσιμες περιπτώσεις και διαφορές, ε, σε άλλες ρυθμίσεις πρόσφατες. Επίσης, να δούμε πώς θα υπάρχει κάποιο δικαστική μόνο απευθυντική θηρίδα. Ένα δικαστήριο να είναι αρμόδιο για τις διατροφές, ένα για επιμέλεια γονική μέρημνα, ένα για ε, διαζύγιο. Οπότε, με τους μηχανισμούς που έχει ο κανισμός σας μέσα στο άρθρο 15 που λέγεται ότι για τη δυνατότητα του να ε, να, να, να, να δοθεί η σκητάλη τη ε, συζήτηση ενό διαζυγίου, μια διαφορά από ένα δικαστήριο στο άλλο, να είναι εύρυθμη αυτή η, η, η συνέχιση της διαδικασίας. Και στα εξεκουάτωρα επίσης να μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα γιατί πάντοτε είναι θέμα της ε, οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Είδαμε τι λέει το άρθρο 24. των ελαχίστων προϋποθέσεων για, την, για να ακουστεί ο ανήλικος σε κάποιες διαφορές Επίση, ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι το να λειτουργεί εύρυθμα η διαδικασία επιστροφής των υλίκων. Τα ασφαλιστικά μέτρα επίση είναι σημαντικά. Εκτέλεση αποφάσεων. Γιατί η εκτέλεση αποφάσεων πολλέ φορέ είναι εθνική υπόθεση και για ζητήματα κοινωνικού δικαίου δεν υπάρχει ικανή πλησίωση. Να, ας πούμε, ε, όσον αφορά την επιστροφή των ελλήνων. Συγγνώμη, έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, αλλά ε, κλείνω. Λοιπόν, το, υπάρχει θέμα τώρα στα πλαίσια του άρθρου 55, θέμα συνεργασίας των εγγονεργών και άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον και αυτή η συνεργασία γίνεται όπως θα έπρεπε, γιατί είναι σημαντική. Επομένω, ε, θα πρέπει να δούμε το πώς και η κοινωνική λειτουργία που βοηθούν τα παιδιά ε, πόσο μπορούν να συμμετάσχουν, να εμπλακούν σε αυτήν την υπόθεση. Άρθρο 56 επίσης. Το έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη τα τέλη του 2014 στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο κάποια άλλα θέματα ανηλίκων που ρυθμίζονται λοιπόν στο άρθρο εκείνο το 56 και όπως ο προηγουμένως η Επιτροπή Γιούγκερ ετώνησε το πόσο προτεραιότητα δίνει στην δικαστική συνεργασία. Είναι πολύ σημαντικός ο κανονισμός 2α για τα θέματα οικογενειακού δικαίου. Οπότε και τώρα προχωρούμε προς την ίδια κατεύθυνση που χαράξαμε. Υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά να κάνουμε σε τεχνικό, τεχνοκρατικό επίπεδο. Πρέπει να γίνει κάποια έκθεση αξιολόγηση. Πρέπει να συνεχιστεί διαβούλευση με ειδικού και εμπειρογνώμονε όπως έχουμε κάνει επανειλημμένα και έτσι να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε εδώ το χρόνο για να σας δεξίσω όλα αυτά. Τονίζω. Είναι πολύ σημαντικό το να ακούμε τη γνώμη σας. Την ακούμε και την προσέχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα. Τώρα θα συζητήσουμε ποιος θέλει να πει κάτι. Κύριε Μαγκίνης, ίσως θέλει να μιλήσει πρώτα. Θα είμαι σύντομη, διότι τα είπα όλα στις εισαγωγικέ παρα... παρατηρήσεις μου. Χαίρομαι που δείχνει ανοιχτό πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε με λογικό τρόπο να ε, ρυθμιστεί τελικά αυτό το ζήτημα. Ως προς τη συνεργασία ανάμεσα στις κεντρικές εθνικές αρχές, ε, όπου και ε, και να γύρει πλάστηκαν, δηλαδή εγκρίνουν ή αποδοκιμάζουν και πού είναι τα προσκόμματα, οι φραγμοί. Κοίταξε, Απαντώντα θα έλεγα πως λειτουργεί σχετικά καλά η συνεργασία ανάμεσα στις κεντρικές αρχές και είναι σε εθνικό επίπεδο προσιλωμένοι, αφοσιωμένοι άνθρωποι που ε, προσπαθούν στις κεντρικές αρχές να εφαρμόσουν ε, αυτές τις αποφάσεις. Όπως λέγαμε, έγγραφο του κυρίου Βανλού, ε, υπάρχουν και κάποια ζητήματα που δεν συζητούνται. Είναι δύσκολη καιρή, χαλεπή καιρή ε, λόγω κρίσης ε, και η έλλειψη πόρων δυσκολεύει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων. Όμως υπάρχει ο μηχανισμός. Αυτό είναι σημαντικό και χρήσιμος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου επίσης. Όντως, είμαστε μια πλατφόρμα συνέβρεσης συζήτησης και όλο και περισσότερο στις έξι περίπου συνεδρίες που έχουμε το χρόνο προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ως φόρουμ, χρήσιμο φόρουμ, ένας διάβλος επικοινωνίας για τις συζητήσεις, παραδείγματος χάρη ε, αφιερώνουμε και χρόνο ε, και για τις διμερείς επαφές ε, πέρα από τις πολυμερείς συσκέψεις. 40 ε, υποθέσεις 40 μεμονωμένες υποθέσεις συζητήθηκαν σε τέτοιες διμερείς επαφές. Νομίζω ότι όλοι κρίνουν είναι χρήσιμο για ε, να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο τις ε, δυσκολίες. Φυσικά οι κεντρικές αρχές συνεργάζονται και εκτός αυτών των συσκέψεων. Όμως παρόλα αυτά όλοι το θεωρούν χρήσιμο. Ευχαριστώ. Τσάρκη λέγομαι. Εκπροσωπώ το ΕΛΚΑ στην Επιτροπή Αναφορών. Η κυρία Μετσόλα, η διακεκριμένη ο απλουστικόλογο δεν μπορεί να παρευρεθεί. Ε, έχει συντάξει την ε, θέση μας και θα ήθελα να την παρουσιάσω. Ε, βάσει τη εμπειρία από την Επιτροπή Αναφορών. Λοιπόν, για τα παιδιά, αναφορές για τα παιδιά ε, σε περίπτωση απαγωγής ε, διασυνοριακής ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε μία αναφορά επίσης ένα διαβατήριο για ταξίδι προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ο ετών ε, ένας γονέας ο οποίος είχε δικαίωμα επίσκεψης ε, για να ε, βλέπει το παιδί του σε ένα κράτος μέλος δεν είχε τα ίδια δικαιώματα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Σχεδόν σε όλες αυτές τις υποθέσεις δεν μπορούσε να αναλάβει οποιοδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο ένδικο μέσο διότι δεν παραβιαζόταν καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι κάποιε εθνική αρμοδιότητα αυτό το ζήτημα. Τα ταξιδιωτικά έγγραφα, παραδείγματο χάρη, ή ε, όταν είχε απειχθεί το παιδί προ μία χώρα που ε, δεν ε, έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τη διεθνή διάσταση των ζητημάτων απαγωγή παιδιών. Ε, υπάρχουν επίσης χώρε που δεν συμμετέχουν στις διατάξεις του Σέγγεν. Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Σέγγεν ε, και άρα ε, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν ε, γίνεται σεβαστό πάντα το δικαίωμα του παιδιού. Μια προσπάθεια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με έναν ασυνόδευτο ανήλικα βλέπουμε ότι είναι εφαρμοστή ο κανονισμός για την προστασία των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και σε περιπτώσει απαγωγή παιδιών, όπου ε, οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωση για τη διαφύλαξη των ε, δικαιωμάτων των παιδιών κατά απαγωγής ε, και κατά εμπορίας εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και σε κράτη-μέλη που δεν ε, ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Υπάρχουν και διάφορα άλλα ε, μέτρα που μπορούμε να επεξεργαστούμε. Παραδείγματο χάρη, αποφάσεις για γονική επιμέλεια και μέλη και δικαιώματα επίσκεψης μπορούν ε, να ληφθούν σε ένα κράτος και να ε, εφαρμοστούν, να εκτελεστούν σε άλλο κράτος βάσει του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Η εκτέλεση γίνεται βάσει εθνικών διατάξεων. Ο στόχος του κανονισμού είναι να εναρμονίσει διαφορετικές εθνικές διατάξεις, ούτως ώστε ευκολότερα να μπορέσουν να επιτύχουν αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος από αυτό ε, τη διαμονή διαμονής τους. Ε, ένα με άλλη πτυχή του κανονισμού Βρυξέλλες 2 είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα ζητήματα που θέτουν οι ετούντες που έχουμε προσφύγει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επιστρέψει την προσοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με ε, ε, τι διασυνοριακέ απαγωγέ. Επίση, η αυξανόμενη κινητικότητα των πολιτών έχει οδηγήσει σε περισσότερε υποθέσει απαγωγή. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλε οι νομικέ υποχρεώσει των επικών των κρατών μελών αναγνωρίζονται και σε λοιπούς πολίτες ε, Παραδείγματος χάρη, κατά τη διάρκεια δικαστικής ε, διαδικασίας, ε, προσφορά βοήθειας ε, στη μητρική τους γλώσσα. Ευχαριστούμε. Κυρία Στάινακα από την Αυστρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις και για το input για ένα πολύ ευρύ θεμάτων σήμερα το απόγευμα. θα ήθελα εν συντομία να στραφώ στο θέμα της διαμεσολάβησης σε θέματα οικογενειακών ζητημάτων και δικαστικών διαδικασιών. Γιατί ο συνάδελφος από αριστερά μου μου δημιούργησε μια, ένα ερώτημα. Μιλήσατε για την δεσμευτική φύση του αποτελέσματος μιας επιτυχημένης διαμεσολάβησης. Εμείς στην Αυστρία συζητάμε συχνά το θέμα αυτό τη διαμεσολάβηση για οικογενειακά ζητήματα και θεωρούμε ότι είναι πολύ ευκταίο για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Αυτό που θα με ενδιαφέρει να μου πείτε είναι το εξή. Ο συνάδελφο, αλλά και εσείς, ε, κύριε Λιβαδόπουλε, να μα μιλήσετε για τη δεσμευτικότητα αυτή τη δικαστική απόφαση. Αυτή η συνθήκη, αυτή η απόφαση πηγαίνει στο δικαστήριο και αποφαίνεται το δικαστήριο μετά. Ή πρόκειται για μια κυκλική διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποιες είναι και οι προθεσμίες για το αποτέλεσμα. Στην Αυστρία έχουμε τη συζήτηση την εξή, γιατί στην παρούσα φάση είναι αθλαντική η διαμεσολάβηση. Υπάρχουν κάπου όμω δεσμευτικοί χαρακτήρε. Και τι γίνεται και με το κόστο για την διαμεσολάβηση. Στοιχίζει χρήματα και στην Αυστρία δεν μπορούμε να το πληρώσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να είναι υποχρεωτικό αυτό, ιδιαίτερα σε οικογενειακέ καταστάσει. Φυσικά Χρειάζονται χρήματα για να υπάρχει καλή πρόσβαση στο δίκαιο. Τι γίνεται όμω στι άλλε χώρε, θα με ενδιαφέρει να το ακούσω αυτό. Σα ευχαριστώ. Και κύριε Λιβαδοπλού. Σα ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Ε. Σε ό,τι αφορά το κατά πόσον ε, μπορούν να επιβληθούν ε, τα αποτελέσματα της Συμφωνίας της Δεμεσολάβησης. Όπως είπα και προηγουμένως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009-52. Η οδηγία αυτή έχει εφαρμοστεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Όλα λοιπόν τα κράτη έχουν βρει τρόπους για να καταστήσουν το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης εφαρμοστέων. Να σας πω τι γίνεται για την Ελλάδα. Πώς εφαρμόζεται το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης. Η συμφωνία η οποία, στην οποία καταλήγουν τα μέρη κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Και από εκείνη τη στιγμή και πέρα επικυρώνονται από το δικαστηρίο και από εκεί και πέρα λοιπόν είναι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο εφαρμοστέα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λοιπόν αναφορικά με την οδηγία αυτή ορίζει το πώς θα εφαρμόσετε στα διάφορα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το θέμα του κόστους τώρα. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Ασφαλώς κάποιες ε, κεντρικές αρχές προωθούν την διαμεσολάβηση. Αλλά πάντα τίθεται το θέμα του κόστους. Αν τα μέρη έχουν τα χρήματα να πληρώσουν την διαμεσολάβηση, αν όχι λαμβάνουν κάποια αρρωγή ενδεχομένω ή μπορεί και όχι από το κράτος και να παραδεχτώ ότι σε πολλές ε, περιπτώσεις το κόστος αποτελεί πρόβλημα για τα μέρη, για το ζευγάρι δηλαδή. Αυτό ασφαλώς εξαρτάται από την εκάστοτε δικαιοδοσία. Ξέρω ότι σε κάποια κράτη υπάρχει κάποια αρρωγή για τέτοιου είδους διαμεσολάβηση από πλευράς του δικού μου κράτους δεν δίδεται χρηματική βοήθεια για τέτοιου είδους διαμεσολάβηση και γενικά για τη διαμεσολάβηση. Αλλά πιστεύω ότι από αυτού θα πρέπει να αποφασίσουμε. Έχετε δίκιο. Ε, ελπίζω να απάντησα στα ερωτήματά σας. Θέλετε κάτι άλλο? Μήπως ξέχασα κάτι? Okay. Uh, uh, Υπάρχουν άλλα σχόλια. If I just may add... να προσθέσω κάτι, γιατί πάρα πολύ σωστά ε, εκτέθηκαν τα θέματα της Επιτροπής Αναφορών όπου είχαμε κάποιες ε, ε, υποθέσεις συγκεκριμένες και σε πολλές περιπτώσεις ε, ήταν πρόβλημα με τα κράτη-μέλη το παράπονο και όχι απλώς ζητήματα ε, διάστασης ή διαζυγίου δικαιώματα ανηλίκων. Θέμα εργασίας αρχών ουσιαστικά προβλήματα στη, σε διάφορα κράτη-μέλη. Και πολλές φορές είναι πάγια αυτά τα προβλήματα, συνεχώς ανακύπτουν. Ε, τελικά είναι εθνική αρμοδιότητα αυτά τα ζητήματα, οπότε είναι δύσκολο ο πολίτης να καταλάβει τι, πώς λειτουργεί το θέμα, τη σχέση ένωσης κράτου μέλους. Επομένως, ε, πάντοτε η ενημέρωση σχετικά με αυτά βοηθάει. Κύριε Σότερ, έχετε πρώτο το λόγο. Σότερ. Ξέρω δεν σας ε, κάλυψε 100% αλλά οπωσδήποτε και θέλω να σας επισημάνω ότι βεβαίως και λαμβάνετε υπόψη βάσει της εμπειρίας μας. Όλα αυτά που λέει ο κόσμος μας, τις τόσες αποστολές, τόσες επιστολές. Όλα αυτές οι επιστολές φτάνουν και στην Επιτροπή των Αναφορών και βεβαίως προσεκτικά εξετάζουμε τις περιπτώσεις αυτές. Δεν μπορώ να συζητήσω κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις τώρα, αλλά πολλές φορές είναι εκτός θέματος οι υποθέσεις κάποιων οι οποίοι βέβαια βρίσκονται πολύ στριμωγμένοι και γι' αυτό τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι συμβαίνει. Πολλές φορές δεν θέλουν να καταλάβουν γιατί εναγωνίως ψάχνουν για κάποια λύση. Λύση που την έχουν αρνηθεί κάπου και την ψάχνουν κάπου αλλού και βέβαια έχουμε κάποια εκπαιδευτική σχεδόν αποστολή για το πού ισχύει το κοινωτικό δίκαιο και πού όχι. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών βάσει του δικτύου βεβαίως και το δίκτυο αποδίδει και λειτουργεί εκεί που ισχύει και που εφαρμόζεται το κοινωτικό δίκαιο. Οπότε και εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορέσουμε για να βοηθήσουμε και εσά και την Επιτροπή Αναφορών για να είσαστε και εσείς όσο γίνεται περισσότερο διδακτικοί. Αλλά πάντως πολλές φορές έχουμε υποθέσεις όπου το πρόβλημα δεν επιδέχεται λύση μέσω του κοινοτικού δικαίου. Δεν βοηθούμε τον κόσμο να προσέλθουν τα πράγματα, ότι έχουν αλλιώς από ό,τι πραγματικά είναι. Πρετέλη. Και έχουμε κάνει μια σχετική ανάλυση για να δούμε το πώς λειτουργούν οι κεντρικές αρχές. Για κοιτάξτε σε 50 ας πούμε της μελέτης μας, εκεί μπορείτε να ένα γράφημα. Εκεί αυτή η κρατική παράσταση λέει ότι σε Αγγλία και Ουαλία υπάρχει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αιτήσεων το οποίο δεν εξηγείται μόνο δημογραφικά. Όμως, αν ρίξετε μια ματιά στο πώς λειτουργούν οι αρχές σε Αγγλία και Ουαλία, θα δείτε ότι εκεί λειτουργούν εύρυθμα αυτές οι υπηρεσίες. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε ούτε στοιχεία να λάβουμε από τις αρχές. μπορούμε καν να βρούμε κάποιο συνομιλητή συγκεκριμένο. Οπότε σε σχέση με αυτό μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ανισορροπίες μέσα στην Ευρώπη. Μπορώ κάτι να προσθέσω, Ελγής Βιαδόπουλος. Δύο λεπτά να απαντήσω σε αυτό που η κυρία Στέναγκερ όσον αφορά την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης. Η οδηγία ορίζει ότι οι δικαστές καλούν τους διαδίκους ενώπιον του διαμεσολαβητή. Πολλές φορές διαμεσολάβηση γίνεται από τον ίδιο τον δικαστή. Αλλά δεν είναι υποχρεωτική τέτοιου διαμεσολάβηση για τέτοιου είδου διαφορέ. Α, ναι, τότε σα ρωτήσω εγώ. Αν είναι υποχρεωτική η διαμεσολάβηση, είναι μια καλή λύση αυτό ή όχι, λέει κύριε Αντελβό. Λιβαδόπουλο. Για κατά τη γνώμη μου, όχι σε τέτοιε περιπτώσει. Δεν είναι καλό να είναι υποχρεωτική η διαμεσολάβηση. Σαφής η απάντησή σας. Ευχαριστώ. Οπότε ολοκληρώσαμε αυτό το πρώτο τμήμα της απογευματινής μας συνεδρίασης. Και τώρα συνεχίζουμε. Θα δώσουμε το λόγο στον ε, καθηγητή Λαγκάρντ από το Παρί Α, το Πανεπιστήμιο το θέμα του είναι το δίκαιο της ονοματοδοσίας και κατά πόσο χρειάζεται να υπάρχει σχετική νομοθεσία. Ah, voilà. Oui, je voudrais dire que je suis très honoré d'avoir été invité par le Parlement européen à exposer mon point de vue. Ευχαριστώ που με καλέσατε να σας πω τις απόψεις μου όσον αφορά το κατά πόσον είναι σωστό να υπάρχει μια νομοθεσία, ονοματοδοσία στην Ευρώπη. Πρώτα πρώτα να σας πω γιατί ανακύπτει το πρόβλημα, ποιοι είναι οι λόγοι και ποιες είναι οι δυνατές λύσεις. Γιατί επομένως ανακύπτει το πρόβλημα, διότι εδώ και κάποια χρόνια προέκυψε το ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και κυκλοφορίας και ως φραγμός αυτό το δικαίωμα προκύπτει το ότι θα πρέπει στην χώρα προορισμού να έχουν διαφορετικό όνομα από το όνομα το οποίο έχουν στην ε, χώρα προέλευσης. Ε, Για κοιτάξτε, έχουμε ας πούμε ένα γαλλογερμανικό ζευγάρι. Γερμανός με Γαλλίδα. Έχει ως τόπο διαμονής την ε, Γερμανία μετά το γάμο, σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, επιλέγουν ένα οικογενειακό επίθετο κοινό και υποθέτω ότι είναι το επίθετο του συζύγου. Οπότε αυτό γίνεται το κοινό επίθετο. Δεν με ακούτε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα επικοινωνία. Δεν λέω. Όχι, αλλά νομίζω ότι ε, ξεπλάγησαν οι κύριε στην αίθουσα που είπατε ότι θα είναι το όνομα του συζύγου. Surprise, madame, mais dans, dans είπα ότι, είπα, είπα ότι ήταν η επιλογή του ζευγού. Οπότε, σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, το πατρόνιμο ε, χάνεται. Οπότε, ε, διαλέγουν το καινούριο επίθετο και όμως στο γαλλικό δίκαιο παραμένει, παραμένει το, το πατρόνιμο. Ακριβώς αυτό το για να καθυσιαστείτε. Οπότε τώρα ε, έχουμε την υπόθεση Γκρούνκιν Πολ. Την διαβόητη. Οπότε είχαμε ένα ανήλικο Γερμανό ο οποίος ζούσε στην Δανία με τους γονείς του. Είχε ένα επίθετο που του δόθηκε από τις Δανικές αρχές, διπλό επίθετο, ε, που ήταν τα δύο επίθετα των δύο γονέων θέλησαν οι γονείς ε, να γράψουν το παιδί στο ληξιαρχείο. Αλλά η, σύμφωνα με τη Γερμανία, ε, σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, δεν μπορεί να έχει διπλό επίθετο το, το παιδί. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενοχλητικά για τους ε, πολίτες. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επανειλημμένα έκρινε ότι και επαγγελματικά και προσωπικά, όλα αυτά είναι πολύ βλαπτικά. Γιατί προκύπτουν έτσι υποψίες, αμφιβολίες, περί την ταυτότητα κλπ. των πολιτών. Επομένως η ρίζα του κακού το ΣΥΠΗΝ είναι οι αποκλίνουσες νομοθεσίες όσον αφορά το ουσιαστικό δίκαιο. Όσον αφορά το αστικό δίκαιο, περί, οι διατάξει περί το επώνυμο. Οπότε, κάποιο έχει ένα επίθετο σε κάποια χώρα. Αυτό όμω μπορεί να είναι το επίθετο του πατέρα ή τη μητέρα. Ή μπορεί να είναι το κοινό επίθετο μετά το γάμο των γονέων. Αλλά σε άλλες χώρες το παιδί μπορεί να έχει ένα σύνθετο διπλό επώνυμο. Πολλές φορές έχουν ε, μεγάλη περιθώρια επιλογής οι γονείς όσον αφορά την επιλογή του επιθέτου του παιδιού. Ε, ε, τώρα, το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο γάμου. Τι γίνεται μετά το γάμο, ο καθένας κρατάει το επίθετό του. Μπορεί ο καθένας να προσθέσει το όνομα του συζύγου του στο δικό του να διαλέξουν ένα κοινό άλλο επίθετο. Να, επομένω, πώ ανεφίσαν αυτά τα προβλήματα, αυτέ τι υποθέσει που σα προανέφερα, αλλά και πολλέ άλλε. Και εδώ πέρα λοιπόν έρχεται το ιδιωτικό διεθνή δίκαιο και λέει ότι το επίθετο είναι θέμα προσωπικό και γνωρίζουμε ότι για πολλά κρατημέλη τα προσωπικά δικαιώματα ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο, αλλά κατά άλλα δίκαια ε, ισχύει το δίκαιο του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής. Στην υπόθεση Γκρουνγκεν Πολ είχαμε απόκληση ρυθμίσεων διότι στην Δανία προβλεπόταν κάτι από το δανέζικο δίκαιο πιο πιο επίσης θα δοθεί. Και έλεγε η Δανία ότι κατησχύει το δίκαιο της κατοικίας, δηλαδή το δανεικό δίκαιο. Ε, αλλά πάλι ε, στη Γερμανία εφαρμοστεί το δίκαιο ήταν το γερμανικό δίκαιο. Άρα πώς θα παρακάμψουμε αυτές τις δυσκολίες και έτσι οι Ευρωπαίοι να μπορούν ανεμπόδιστα πραγματικά να διακινούνται. Πρέπει πρώτα πρώτα να αποκλείσουμε επέμβαση ευρωπαϊκή όσον αφορά το δικαίωμα επιλογής. Γιατί εδώ πέρα ισχύει αρχή της Η ονοματοδοσία τέλος πάντων η επιλογή του επιθέτου είναι κάτι το οποίο προκύπτει από παράδοση, πολιτισμό, κράτους ε, μέλους και η πολυμορφία σημαίνει ότι θα πρέπει η εθνική ταυτότητα και η βιοτυπία να αντικατοπτρίζονται και σε αυτό το επίπεδο. Οπότε εδώ υπάρχει μια ελευθερία των μελών σε αυτά, σε λογικά επίπεδο, όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα πρέπει να ασκείται έτσι, ούτω ώστε να υπάρχει σεβασμό του ιδιωτικού βίου και να μην υπάρχουν ε, δυσμενεί διακρίσει, αλλά μέχρι εκεί. Από την άλλη μεριά όμω, αυτό το οποίο είναι επιθυμητό και δυνατό να παρέμβουμε μέσω του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οπότε σε επίπεδο ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ε, υπάρχουν δύο δρόμοι που να ακολουθήσει το κοινωτικό δίκαιο. Ή μπορεί να γίνει μια ενοποίηση, κωδικοποίηση των κανόνων για την ε, άρση των συγκρούσεων ε, δικαίων και ένας και μόνο κανόνας να ορίζει την επιλογή του επιθέτου σε όλα τα κράτη-μέλη. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι να αναγνωρίζονται ε, στα, σε όλα τα κράτη-μέλη τα επίθετα τα οποία έχουν ε, δοθεί σε άλλο κράτος μέλος. Άρα, αναγνώριση των επιθέτων. Από τη μία μεριά ή από την άλλη κανόνες επίλυση των συγκρούσεων διαφορετικών ρυθμίσεων. Νομίζω ότι παρουσιάζει περιορισμένα πλεονεκτήματα μία τέτοια λύση. Ε, κοιτάξτε τι έγινε με αυτό το γαλλογερμανικό ζευγάρι. Η γυναίκα κράτησε το επιθετό της σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο. Αλλά σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο το, το χάνει και παίρνει το κοινό επίθετο. Αυτό αυτό δεν είναι εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό που είναι εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία είναι το ότι το επίθετο σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο δεν θα αναγνωριστεί στη Γαλλία. Στην υπόθεση Γκρούνγκεν Πολ δεν ήταν το πρόβλημα οι διαφορετικές ρυθμίσεις Δανίας και Γερμανίας αλλά ήταν η άρνηση των γερμανικών αρχών να αναγνωρίσουν το επίστο το οποίο δόθηκε ε, σύνομα στην Δανία. Πάντως θα πρέπει να αναδείξουμε τώρα τον Ολλανδικό του 2011 όπου υπάρχει ρύθμιση ε, εντελεχής σε σχέση με την αναγνώριση των επιθέτων. Θεωρώ ότι η αναγνώριση των επιθέτων θα πρέπει να αφορά και την αλλαγή του επιθέτου. Επί τη βάση κάποιας δήλωσης, κατόπιν ας πούμε ε, γάμου, κατόπιν αλλαγής ε, ε, οικογενικής κατάστασης και επίσης όσον αφορά ονόματα που έχουν δοθεί σε Ευρωπαίο πολίτες σε κάποια τρίτη χώρα. Αναγνώριση σε κράτος μέλος. Και καταχώρηση αυτού του επιθέτου στο ληξιαρχείο της χώρας. Επομένω, πρόκειται για αναγνωρισμένο επίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα πρέπει να γνωριστεί και αλλού. Είναι δύσκολο το θέμα εδώ, γιατί θα πρέπει να δούμε ε, κατά πόσον αυτό του είδου η αναγνώριση έχει να κάνει με κάποιο είδου εξάρτηση από, από εθνικότητα, από ε, ε συνήθι τόπο κατοικία ή επιλογή δήλωση του ίδιου του πολίτη. Είναι πολύ συζήτηση βέβαια το θέμα, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι προϋπόθεση απαραίτητα. Η αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια τέτοια προϋπόθεση η δημόσια αρχή ενώπιον της οποίας α, κρίνεται η υπόθεση θα πρέπει να διαπιστώσει τι γίνεται με το επίθετο. Οπότε και αυτό πρόκειται να αποτελέσει λόγω καθυστέρησης έναν φραγμό στην ελεύθερη κυκλοφορία. Παμπούσε. Ένας κανονισμός να συμπληρώσει την απόφαση της Επιτροπής τη 24η Απριλίου του 2013, όπως όπω είπαμε το πρωί θα μπορούσαμε ε, κατά τον ίδιο τρόπο να το ρυθμίσουμε όπως με την ε, αποδοχή των δημοσίων εγγράφων την ε, αναγνώριση των δημοσίων εγγράφων που προχωρούνται από λαδαπή αρχή. Α, είδατε, ε, τελείωσα λίγα τρόλεπτα λιγότερο από το χρονικό όριο. Σας ευχαριστούμε για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση καθηγητά. Ναι και εγώ στην αρχή κάπως ε, εντυπωσιάστηκα, με ξένησε το θέμα, αλλά δεν είναι ενδιαφέρον το θέμα. Θέλει κάποιος να θέσει ερώτημα. Yes, Mr. Ε, Κύριε Κλέντς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, πολύ μου άρεσε. Και διάβαζα ταυτόχρονα και το έγγραφο και πρόσεξα ότι δεν υπάρχει αναφορά σε αγγλοσαξονικές ε, περιπτώσεις. Ε, τι γίνεται βάσει αεραλυντικής ε, ε, παράδοσης, ε, στη Σκωτία παραδείγματο χάρη. Ε, ή κρατάει το πατρικό της η γυναίκα ε, ή παίρνει το επώνυμο του συζύγου. Και για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας ε, λέγεται η γυναίκα η κυρία Τζόνς ή Σμιθ. Είναι με διαζευτικό. Ε, και σε χώρες common law λοιπόν Ε, ίσως έχετε άλλες ιδέες, παρά δεν είναι αναφέρεστε σε αυτό το ζήτημα στο εγγραφό σας. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν αναφέρθηκα ε, στις χώρες Common Law στη μελέτη μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτές τις χώρες, διότι δεν αρνείστε ποτέ την αναγνώριση ενός ονόματος και δεν δημιουργείται προβλήματα. Στην Διεθνή Επιτροπή Ληξιαρχείων ε, είχα, έχω κάποια εμπειρία ε, γιατί έχουν συνταχθεί διάφορες συμβάσεις για τα ονόματα και η αντιπροσωπή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας ή τουλάχιστον του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί τότε η Ιρλανδία δεν ήταν μέρος μας έλεγε ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα ζητήματα, αλλά υπηρετικά, continental, υπηρετικά. Ευχαριστώ. That just goes to show there are some things which are simple about the... Να λοιπόν, αυτή η απόδειξη το ότι κάποια πράγματα είναι απλούστερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, si, si, je peux, si je peux ajouter... Όχι, μπορώ όντω να προσθέσω κάποια πράγματα ουσιαστικά θα ήταν πάρα πολύ καλό να ήταν όλοι εξίσου φιλελεύθεροι όσο το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεφορείων να αναγνωρίζουν την ονοματοδοσία άλλων κρατών. Σας ευχαριστώ πάντα. Γαλλιστή ο κύριος Κράου. Λοιπόν, με τις ε, φιλοφρονήσεις νομίζω κλείσαμε. Θα σας πρότεινα τώρα να διακόψουμε μέχρι τις 4.30 ή και 20. Ε, καλά, 10 λεπτάκια. Να επιστρέφουμε 3 και 20 για τον τρίτο γύρο. Τι. Oui, c'est euh, incroyable que l'écho s'est dit, a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

I am very sorry to interrupt you, but I propose that we start. Uh, we have to finish at, eight, at six o'clock. Ε, πρέπει να αρχίσουμε για να τελειώσουμε ε, στις 6. Ας μην καθυστερούμε λοιπόν. Για να αρχίσουμε το τρίτο ε, μέρος ε, των συζητήσεών μας θα δώσω το λόγο στον δόκτωρα Χάρμ Σέπελ, καθηγητής οικονομικού δικαίου σχολείου διεθνών σπουδών των Βρυξελών Πανεπιστήμιο του Κέντ στις Βρυξέλλες. Uh, ε, Έχετε το λόγο και ελπίζω να σας ακούν ε, οι παρευρισκόμενοι. Ευχαριστώ. Θα φωνάζω για να με ακούν. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Είναι τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ. Είναι δύσκολο βεβαίως, διότι μου ανέθεσαν να μιλήσω για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο ως εργαλείο για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν είμαι ειδικός, ζητώ συγγνώμη. Um, Λοιπόν, με δύο διαφορετικού τρόπου αναφέρεται κανεί στο ιδιωτικό διεθνέ δίκαιο. Πρώτον, για να αναφερθεί στην ε, αύξηση της σημασίας ε, των ε, ιδιωτικών των φυσικών προσώπων στην παγκόσμια διακυβέρνηση και δεύτερον χρήση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για την διευθέτηση συγκρούσεων ανάμεσα σε διαφορετικές ενόμες τάξεις ή τουλάχιστον για να ρυθμιστεί η διάδραση ανάμεσά του. Υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα. Το ένα σχετίζεται με αυτούς που για λόγους ε, ε, ασφάλειας και υγείας ε, θέτουν τα πρότυπα και το δεύτερο καθεστώς σχετίζεται με επενδυτικές συμβάσεις. Αυτά και τα δύο συστήματα και τα δύο καθεστώτα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η κυβέρνηση. Χρησιμοποιείται δε ως μέσο εξουσιοδότησης ε, η σύμβαση. Τα TBT, τα για τα τεχνικά, δηλαδή τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, χρησιμοποιούνται δεσμευτικά πρότυπα ε, που εγκρίνουν τα ε, κράτη-μέλη Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σε εθνικά διαμεσολαβητικά όργανα για να ρυθμιστούν οι διασυνοριακές διαφορές, από κράτος σε κράτος δηλαδή. Ε, και στις δύο περιπτώσεις δημιουργούνται συγκρούσεις δικαίου και επίσης τίθεται διάφορα ζητήματα των σχέσεων ανάμεσα στις διαφορετικές ένωμες τάξεις, διαφορετικά νομικά καθεστώτα. Στην πρώτη περίπτωση είναι σχετικά απλό αυτό που λέω, ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση δηλαδή προκύπτει από την αλληλεπίδραση ρυθμιστικών τάξεων ε, και οι προσπάθειες προστασίας από τα εθνικά συστήματα είναι τελικά αντιπαραγωγικές ακριβώς όπως και να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα εθνικά οικονομικά και εμπορικά συστήματα από αυτή την ελληνεπίδραση. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο για την ρύθμιση της αλληλεπίδρασης αυτών των διαφορετικών συστημάτων. Ας πάρουμε πρώτα τα διεθνή πρότυπα. Ένα μεγάλο κομμάτι των προτύπων στον τομέα του περιβάλλοντος, το, της κατάρτισης ε, λογαριασμών, ε, της οικονομίας ε, προκύπτουν από συμβάσεις ανάμεσα σε ιδιωτικούς φορείς. Ως προς την εκπόνηση των προτύπων, χρησιμοποιούνται εγχειρίδια επαγγελματικών ενώσεων, πρόκειται για μια επαχθή διοικητική ε, διαδικασία και αναμφίβολα αυτό προέρχεται από αναγνώριση διαφορετικών νομικών διατάξεων από διάφορα κράτη-μέλη. Όσο και να νομιμοποιούνται αυτά τα συστήματα, δεν μπορούν να αποκτήσουν το καθεστώς ε, της νομικής διάταξης, διότι δεν προκύπτουν από μια νομοτεχνική διαδικασία. Όπως ε, συμβαίνει, παραδείγματο χάρη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιπίνε. Ή θεωρούνται αυτά τα πρότυπα μάλλον ως τελεσμένα γεγονότα. Το πρόβλημα είναι ότι ρυθμιστικές απαιτήσει ε, ε, γεγονότων δεν μπορούν να τεθούν ακόμη και αν πρόκειται για νομικής αξίας γεγονότα. Ε, ε μια περίπτωση δικαστηρίου, παραδείγματο χάρη, ήταν κατά ε, μιας επαγγελματικής ένωσης ε, για τις ε, σαρδίν, ε, συγγνώμη, ε, που δεν αναγνωρίστηκαν τα πρότυπα αυτής της ένωσης επειδή δεν συμβάδιζαν με έναν κώδικα του κόντεξ αλιμεντάριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναζητήθηκε μια συνενετική λύση. Αυτό το συγκεκριμένο πρότυπο είχε εγκριθεί στη Ρώμη την Παρασκευή το απόγευμα. Ε, είχαν φύγει οι περισσότεροι ε, και τελικά ε, νεκρύθη το πρότυπο χωρίς τις, τα, τα προβλεπόμενα, προβλεπόμενες διατάξεις, δηλαδή η συμμόρφωση με τον κόντεξ. Τι συνέβη στη συνέχεια. Το πρότυπο κανονικά αναγνωρίζεται όταν εγκρίνεται από έναν διεθνή οργανισμό. Η διαδικαστική ακαιρεότητα, αν θέλει, της διαδικασίας έγκρισης δεν απασχολεί κανέναν κατά τα άλλα. Και πού ήταν το πρόβλημα λοιπόν. Το πρόβλημα ήταν πως το συμπέρασμα δεν είχε ως στόχο να επηρεάσει τις οικίες απαιτήσει των διεθνών προτύπων που έχουν ε, εγκρίνει διεθνείς οργανισμοί στις εγχώριες επιχειρήσεις τους. Δηλαδή, η συμφωνία TBT για τους τεχνικούς φραγμούς υπάγεται σε αυτήν την διεθνή σύμβαση περί θεσπίσεως προτύπων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Διεθνής Οργανισμός δεν πρέπει να αναζητά τη συνενετική λύση για την εκπόνηση των προτύπων. Δεν το αποφασίζουμε εμείς. But it should be. Recently uh, Μετά από τις αρδέλες ε, έχουμε την περίπτωση Μεξικού, είπα, για τον τόνο που ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση για τις ε, σαρδέλες ε, και για τα διεθνή πρότυπα αλλάζουν οι κανόνες και απαιτείται πλέον συνένεση. Αυτό πώς ακριβώς συνέβη Βάσει της σύμβασης ε, της Βιέννης για την ερμηνεία των συμβάσεων ε, ανακηρύχθηκε ως ε, νομικά αναγνωρίσιμη διαδικασία αυτή της εκπόνησης των προτύπων. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο της εξουσιοδότησης φυσικά υπακούν σε κάποιους διαδικαστικούς κανόνες και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Α περάσω στο επόμενο θέμα, στα πλαίσια τη ε, Παγκόσμια διακυβέρνηση. Ε, διαμεσολάβηση ε, ως προς τις επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν τις συναλλαγές σε αυξανόμενο ρυθμό και βλέπουμε πως η διαμεσολάβηση σε εμπορικές υποθέσεις αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς αυτό ήταν αναμενόμενο, όμως ε, η διαμεσολάβηση για τις επενδυτικές συμβάσεις ε, έχει αυξηθεί με ακόμη ταχύτερο ρυθμό και αυτό δεν ήταν αναμενόμενο το 1990. Ε, υπήρξε μια έκρηξη του αριθμού των συμβάσεων και το 2000 ο αριθμός των υποθέσεων ε, επίσης γνώρισε μια έκρηξη ε, των υποθέσεων των οποίων επιλαμβάνονται τα δικαστήρια στην εμπορική διαμεσολάβηση μπλέκεται το διεθνές ε, ιδιωτικό δίκαιο και δεν μπορούμε να βασιστούμε στην αυτονομία ε, των διαδίκων ε, των μερών όπως η εμπορική διαμεσολάβηση. Έχει προταθεί ότι η διαμεσολάβηση είναι θέμα δημοσίου δικαίου, παγκοσμίου αν θέλετε διοικητικού δικαίου και ουχή ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ε, δεν θα ήθελα να πω σε λεπτομέρειες για το επενδυτικό καθεστώς. Υπάρχει ένα ζήτημα που θα ήθελα να σχολιάσω, αλληλεπίδραση με άλλες ένομες τάξεις. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Προβλέπουν οι συμβάσεις κυρίως δύο διαφορετικά είδη προτύπων. Πρότυπο Τη μη διακριτική μεταχείρισης, αυτό είναι σχετικό, και το απόλυτο πρότυπο ε, της ε, μη απαλωτρίωσης ε, χωρίς αποζημίωση, καθώς και το ΦΕΤ του, της ισότιμης δηλαδή και δίκαιη μεταχείριση. Παραδοσιακά η πρώτη διαδικασία το όταν ο επενδυτής, αλλοδαπός επενδυτής, λειτουργούσε με τρόπο που παραβίαζε τα διεθνή πρότυπα ανεξαρτήτως υπηκότητος ε, του επενδυτή. Παρ' αυτά, με την μεταξέλιξη του επενδυτικού δικαίου, αυτό το πρότυπο ΦΕΤ ε, υπερεύει αυτά τα όρια για την δίκαιη μεταχείριση και έτσι η χώρα υποδοχής υποχρεούται να διατηρεί ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Όπερ μα οδηγεί στο ότι τα μεσολαβητικά δικαστήρια για να πληρούν αυτές τις υποχρεώσεις διεθνούς δικαίου ζητούν από τους αλλοδαπούς επενδυτές να μην γύρουν υποθέσεις σε περιπτώσεις όπου δεν θα το έκαναν οι επενδυτέ δηλαδή συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις. Θεωρητικά υπάρχουν και τα δικαιώματα συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία επιπροσθέτως οπότε ε, το εθνικό δίκαιο προστατεύει όσους δεν έχουν άλλα μέσα, άλλους τρόπους ε, να επηρεάσουν ε, ε, με τις πολιτικές παραδείγματος χάρη διασυνδέσεις τους τις εξελίξεις στην υπόθεσή τους. Τα κράτη-μέλη φυσικά διατηρούν ακέραιο το δικαίωμά τους να νομοθετούν για το κοινό συμφέρον για το καλό της δημόσιας τάξης. Στην υπόθεση Γιούκος, παραδείγματος χάρη, το δικαστήριο έπρεπε να εξηγήσει ε, κάτι σχετικά επώδυνο. Ε, έφτασε η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, που αποφάσισε ότι δεν υπήρξε μια παραβία στο άρθρο 1 πρωτόκολλο 1 της Σύμβασης δηλαδή για τα περιουσιακά δικαιώματα και έπρεπε το δικαστήριο να εξηγήσει γιατί οι επενδυτικές συμβάσεις προστατεύουν καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών παρότι τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Υπάρχουν ελάχιστα δικαιώματα που κατοχυρώνονται ανεξαρτήτως της βούλησης ε, του ε, ατόμου και βάσει αυτών των συμβάσεων υπάρχουν ξεκάθαρες ε, διατάξεις που παροτρύνουν τους επενδυτές να δραστηριοποιούνται βάσει αυτών των δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει πως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται το περιθώριο ερμηνείας για να αποδυναμωθούν αυτά τα δικαιώματα όπως παραδείγματο χάρη στις συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η... Τα πρότυπα προστασίας ε, των επενδυτών ε, είναι υψηλότερα σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, Ζητώ συγγνώμη, αλλά μπορείτε να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα. Σχεδόν έφτασα, πρόεδρε. Εάν ένα δικαστήριο επιληφθεί της απόφασης, ε, θα αναγνωρίσει ότι ε, ένας αλλοδαπός επενδυτής ε, δεν μπορεί να εγείρει μία αξίωση ε, αν δεν θα το είχε πράξει και ένας εγχώριος επενδυτής βάση της νομοθεσίας για την προστασία των επενδυτών και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμπέρασμα θα είναι απλό. Τα Δικαστήρια διαμεσολάβησης θα πρέπει να προστατεύονται από την πολιτική επιρροή και η αυτονομία αυτή όμως σε σχέση με το οικείο εθνικό δίκαιο και το δίκαιο διαμεσολάβησης δεν αποτελεί παρόλα αυτά εχέγγυο. Σας ευχαριστούμε δόκτωρα Σόπελ. Καλωσορίζω τον δόκτωρα Παύλο Κόρτες από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ για το επόμενο ε, σημείο για τη διαδικασία ανάκτησης ε, μικρόπωσων αξιώσεων. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που συμμετέχω εδώ στη ζήτηση της Επιτροπής σας για να σας παρουσιάσω αυτή την μελέτη που αφορά τη διαδικασία μικροδιαφορών. Αυτή η διαδικασία είναι εκούσια, μη υποχρεωτική για διασυνολογικές μικροδιαφορές μέχρι τα 2.000 ευρώ. σε εξαιρετικές περιστάσεις ε, καταφύγει κανείς αυτό. Και υπάρχουν συγκεκριμένες σύντομες προθεσμίες. Δεν είναι υποχρεωτικό να παρίσταται συνήγορος, πάντως ε, το 30% των διαδίκων προτιμά να έχει. και η τελική απόφαση είναι εκτελεστή χωρίς να χρειάζεται δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει το εκτελεστό της αλλοδαπής απόφασης. Γενικώ, αυτή η διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική από τις εθνικές διαδικασίες για τις διασυνορικές διαφορές. Πάντως, στην πράξη δεν χρησιμοποιείται και πολύ. Έχουμε μόνο 100 υποθέσεις ανά κράτος δηλαδή, περίπου συνολικά περί τις 3.000. Ε, Έχουμε συντάξει μια σειρά μελετών και θα υποβάλουμε κάποια πρόταση, ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται για διάφορα προβλήματα όπως την μη χρήση της διαδικασίας. Ίσως ο κόσμος δεν είναι τόσο ενημερωμένος, δεν την ξέρει τη διαδικασία και από το κέντρο καταναλωτών πρόκειψε ότι μόνο 12% των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία. Αλλά προβληματίζει περισσότερο το ότι 53% των δικαστών δεν γνωρίζουν την διαδικασία που είναι αυτοί που την διαχειρίζονται. Επίσης, προέκυψε ότι πολλές φορές θεωρούν ότι δεν, είναι τόσο, δεν έχουν τόσο διαφάνεια ε, τα έξοδα, τα δικαστικά που σε πάγει αυτή η διαδικασία. Ούτε επίσης είναι τόσο σαφές ποιοι καλύπτονται αυτή τη διαδικασία. Ε, αυτό ξεκίνησε για καταναλωτές και για επιχειρήσεις, αλλά στην πράξη βασικά κάποιες επιχειρήσεις ή κάποιοι πολύ μορφωμένοι καλύπτονται από μια τέτοια διαδικασία. Πολύ, πολύ λίγοι δηλαδή. Γιατί η... με τον λόγο δεν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την εκτελεστότητα που εξασφαλίζεται μέσω του εθνικού δικαίου. Εάν είχαν πάει στις εθνικές αρχές οι καταναλωτές, θα είχαν μεγάλα προβλήματα. Οπότε θα πρέπει να πάνε σε άλλο κράτος μέλος, με άλλη διαδικασία, για να πετύχουν την ίδια δουλειά. Άρα, οι ενός καταναλωτών δεν ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διαδικασία και θεωρούν ότι η βασική δυσκολία για να χρησιμοποιηθεί ε, αυτή η διαδικασία των μικροδιαφόρων είναι το ζήτημα του πώς θα εκτελεστεί η απόφαση. Έχουμε υποβάλει μια σειρά προτάσεων. Αυτά δημοσιεύτηκαν στις 19 Νοεμβρίου του 2013. Χαιρετίστηκε με επιτυχία η πρότασή μας. Είχαμε προτάσει και για να διευκολυνθεί η διαδικασία της εκτέλεσης απόφασης, διαταγή πληρωμής, πώς θα παραγαμφθούν οι αντιρρήσεις του διαδίκου. Ρυθμίση του ποσού. Όταν έχουμε κάποια αξίωση περίπου τα 5.000 ευρώ, τότε αυτό φτάνει περίπου το ύψος του δικαστικών ε, εξόδων όταν κανείς έχει αξίωση 10.000 ευρώ. Επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το τι θεωρείται ο ορισμός του τι θεωρείται διασυνοριακή διαφορά. Επίσης η ηλεκτρονική επικοινωνία για να υπάρχουν κάποιου είδους, ε, είδους προφορικές τέλος πάντων διαδικασίες και σε σχέση με τα δικαστικά έξοδα. Γιατί είπαμε ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχει μια διαδικασία στα τοπικά δικαστήρια. Αυτό θα ανέβαζε τις δικαστικές δαπάνες θα ήταν πιο οικονομικό εάν υπήρχε ένα μόνο δικαστήριο το οποίο θα συνδύαζε την χρήση της τεχνολογίας αλλά και την διοικητική ούτως υπήν διεκπαιρέωση της ε, υπόθεσης και έτσι θα είχαμε κάτι σαν οικονομία κλίμακας. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα πρέπει να πάνε στο 10% το ποσό των, ε, των δικαστικών εξόδων. Αυτό ξέρουμε θα, είναι, θα προκαλέσει διαφωνία στα κρατημέλη. γιατί α πούμε στα 10.000 ευρώ πάμε στα 1.000 ευρώ έξοδα που είναι πολλά. Ε, είπαμε πάει πάνω από τα 2.000 να είναι 5% τα έξοδα. Επίσης έχουμε προτείνει η μετάφραση του κλειστού τίτλου να αφορά μόνο το διατακτικό. Επίσης, βοηθήσαν το κατημέρι σε κάποιες απορίες που είχαν, αλλά δεν ξεκαθαρίστηκε το εξή. Τι γίνεται με κάποιον ο οποίος θέλει να γύρει αξίσου σε άλλο κράτος μέλος. Και εκεί να είναι το αρμόδιο δικαστήριο. Κατά γνώμη μου, το προβληματικό σημείο είναι ότι όταν τα οι διάδικοι θέλουν να δοθεί μια λύση θα πρέπει να γίνεται μια συζήτηση. Πάντως οι περισσότερες προτάσεις που έχουν γίνει είναι θετικές, αλλά θα πρέπει να συμπληρωθούν. Πρώτα πρώτα όπως είπαμε πριν, για να διευκολυνθεί η εκτέλεση. αλλά δεν αρκεί η ενημέρωση των χρηστών για το σε ποιο website θα πρέπει να πάνε, αλλά θα πρέπει να, να τους ξεκαθαριστεί ότι θα γίνει ε, η εκτέλεση απόφαση με μια διαφορετική διαδικασία και σε μια άλλη διαφορά, σε μια άλλη χώρα. Γιατί αυτό οδηγεί σε κάποια έξοδα τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μόνο ε, μπορεί να τα ανακτήσει ο διάδικος. Άλλη μας πρόταση. Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση για αυτή τη διαδικασία μικροδιαφορών. θα πρέπει να συσχετιστεί η διαδικασία με τη διαδικασία δημεσολάβησης. Είπαμε ότι θα έχουμε την πλατφόρμα επιλυση διαφορών μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 και εκεί θα καλύπτουμε καταγγελίες καταναλωτών για διαφορές που προκύπτουν από ηλεκτρονικό εμπόριο και όταν δεν είναι το να γίνει επίλυση αυτών των διαφορών τότε οι διάδικοι θα πρέπει να πηγαίνουν στο αρμόδιο δικαστήριο για να επιλύσουν αυτή τη διαφορά. Και να ισχύει αυτή η διαδικασία μικροδιαφορών. Θα πρέπει να επισημαίνεται κάθε φορά από τους διαδίκουσαν αν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει αυτή τη ε, διαδικασία ή αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ε, διαμεσολάβηση. Κάποιε χώρε όπω η Ιρλανδία έχουν χωρε οπως η ιρλανδια διαδικασία και έχουν επομένως ε, τα, δικαστήρια μια τέτοια εξοικείωση και υπάρχει κάποιο διαμεσολαβητή ο οποίος διαπραγματεύεται και, και τηλεφωνικά με τα δύο μέρη. και σε πολλές περιπτώσεις, περισσότερε περιπτώσει, καταλήγουν σε συμβασμό οι διάδικοι πριν την εκδίκαση της απόφαση. Όμως τώρα μιλούμε για τα διασυνοριακά. Άρα μέσω ενός κανονισμού θα πρέπει να καλύπτονται και οι διασυνοριακές διαφορές. Και οι ενώσει καταναλωτών επίσης ε, μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν διαδίκους ιδίω από γλωσσικής πλευράς. Παρακαλώ, καταλήξτε κάπου. Ναι, ολοκληρώνω και σας τονίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι πανάκια η διαμεσολάβηση, αλλά είναι έχει καλύτερη σχέση κόστος αποτελέσματος και, και ικανοποιεί πολύ περισσότερο από την ένδικη πλήση των διαφόρων. Και έτσι δημιουργείται περισσότερη εμπιστοσύνη προς το σύστημα βουλουράς των καταναλωτών για τέτοιες διασυνορικές διαφορές. Ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στον συναδελφό μου, την ε, κυρία αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ε, Γιούρι, την κυρία Λίτιγκα και η οποία είναι και η συγγήτρια για την αναθεώρηση του κανονισμού περί μικρών διαφορών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσω στα πολωνικά, μια και όλα μου τα έγγραφα είναι προετοιμασμένα σε αυτή τη γλώσσα. Να ευχαριστήσω όμω ε, πολύ του ομιλητέ για την εισαγωγή τώρα να κάνω κάποια σχόλια και ελπίζω στη συνέχεια να είναι καρποφόρα η συζήτησή σας. Ε, να ξεκινήσουμε με το θέμα του ονόματος του κανονισμού αυτού. Ήδη από εκεί είχαμε κάποιες αμφιβολίες. Κατά πόσον θα έπρεπε να μιλάμε για μικροδιάφορες, γιατί μικροδιάφορες αυτό σε κάθε χώρα μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό. Εν γέννη, θα θέλαμε το εργαλείο αυτό να είναι ελαφρύ, κατανοητό και να λειτουργεί σωστά. Για όλες τις αξιώσεις μέχρι 10.000 ευρώ. Αξιώσεις μέχρι δε, το ποσό αυτό. Δεν μας αρέσει τόσο πολύ η όρος ε, μικροδιόφορων Στη Λιθουανία, στη Βουλγαρία δεν είναι μικρά τα ποσά αυτά, ξέρετε. Σε σχέση με τους μισθούς. Στην Βουλγαρία και στη Λιθουανία αντίστοιχα. Στην Επιτροπή λοιπόν ε, Γιουρί Νομικών Υποθέσεων υπάρχει γενικά συμφωνία και συνένεση ότι αυτό το εργαλείο θα έπρεπε να λειτουργεί καλύτερα και θα πρέπει να προωθηθεί όχι μόνο μεταξύ των ε, καταναλωτών, αλλά και μεταξύ των δικαστών. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε, γιατί η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρασε από μεγάλη ανάλυση. Θα ήθελα παρόλα αυτά να αναφερθώ σε κάποιε λεπτομέρειε που κάνουν τη ζωή του καταναλωτή πιο δύσκολη. Τα δικαστικά τέλη. Δεν μπορεί κανεί να τα πληρώσει με πιστοτική κάρτα. Οι πληρωμές αυτές πρέπει να γίνουν μέσα στο δικαστήριο. Θέλουμε λοιπόν τα τέλη αυτά να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται, προκειμένου ο πολίτης να μην υποθαρρύνεται όταν πρόκειται για διαφορές ε, χαμηλών ποσών. Αυτή η αξίωση στην ευρωπαϊκή αγορά οδήγησε στην εξή κατάσταση. Οι καταναλωτές τελικά δεν τυχάνουν καλή ε, αντιμετώπιση ε, και τελικά δεν αρκεί αυτή η αντιμετώπιση. Τώρα λοιπόν ανοίξουμε τη συζήτηση. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Ο κύριος Μπούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ εκτιμώ αυτά που ακούσαμε και από τον καθηγητά και από την... τους συναδέλφους. Εκτιμώ και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά παράλληλα πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε... Ακουγόμαστε. Είχαμε λοιπόν αυτές τις αξιώσεις ε, μέχρι 10.000 ευρώ την, ε, μέχρι 2.000 ευρώ. Τώρα συζητάμε κατά πόσο αυτό θα πρέπει να φτάσει στα 10.000 ευρώ. Στην ε, ομάδα μου, στο ΕΛΚ, συζητάμε μήπως θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 2.000 ευρώ για τις ιδιώτες και 10.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι χρειάζεται αυτή η ρύθμιση στο αστικό δίκαιο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Είναι πολύ σημαντική για τον πολίτη, αλλά παράλληλα αποτελεί και μέτρο πρόληψης τέτοιων ε, περιπτώσεων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το σημείο αυτό, μην το ξεχνάμε, γιατί αν αυτοί που συμμετέχουν, αν οι φορείς στην κοινωνία ξέρουν ότι υπάρχει ένα απλό και εύστοχο εργαλείο που λειτουργεί τόσο καλά, σίγουρα θα υπάρχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον προκειμένου όλοι να τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα πιο συγκεκριμένα μιλώντας και για το πεδίο εφαρμογή της διαδικασία αυτής. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη λογική αυτή. Είτε μιλάμε για 2.000, 5.000, 10.000 ευρώ. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να κάνουμε το εξή. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να το αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούνται και στο εργασιακό δίκαιο, όταν πρόκειται για μια εργασιακή σύμβαση, μια μεμονωμένη εργασιακή σύμβαση. Να ισχύουν αυτά λοιπόν και σε αυτόν τον τομέα. Και εδώ λοιπόν μιλάω για αποζημιώσεις, αμοιβέ. όχι για ε, αμοιβέ αποζημιώσεις. Αν υπάρχει μια μεμονωμένη διαδικασία. Θα πρέπει να ισχύει αυτό το εργαλείο. Έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια πολίτες αυτή τη στιγμή και πιο πολλού μην σα πω που ζουν σε μια άλλη χώρα εκτός τη πατρίδα τους και δουλεύουν εκεί. Υπάρχουν λοιπόν πολλές καταστάσεις και πολλές περιπτώσει όπου έχουν συνάψει μια ατομική εργασιακή σύμβαση και η εργασιακή αυτή η σύμβαση καταγγέλλεται χωρίς να πληρώνεται ένα μισθός για παράδειγμα. Δεν έχει ο πολίτης ε, για παράδειγμα χρήματα για να καταγγείλει αυτή την ε, παραβίαση και αναγκάζεται να επιστρέψει στην ε, πατρίδα του. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα να μπορεί στην πατρίδα του να καταγγείλει την εκάστοτε εταιρεία, γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει οποιαδήποτε λύση στην παρούσα φάση για το πρόβλημα αυτό. Αν η εκάστοτε εταιρεία, για παράδειγμα, έχει αντιπροσωπεία στη χώρα του εργαζόμενου, τότε ναι, μπορεί να δράσει. Αν όχι, δεν μπορεί να αντιδράσει. Λοιπόν, να το σκεφτεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι χρειάζονται επιπρόσθετα εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πραγματικά τον πολίτη, προκειμένου να έχει μια, πραγματικά, μια πραγματική ευκαιρία για πια απλή ζωή. Για του διάφορου δασμού, τέλη, φορολογίε κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο αυτό εδώ, γιατί συνήθω πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσει που δεν έχουν πολλά χρήματα. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά η πληρωμή, όχι απαραίτητα μέσα στα κτίρια της υπηρεσίας, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να σηκωθεί και να πάει εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει άνετα σε μια τράπεζα και να αποστείλει μετά ταχυδρομικά την ε, απόδειξη πληρωμής. Δεν ξέρω, λέω τώρα ένα παράδειγμα αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον Ευρωπαίο πολίτη και νομίζω ότι αυτό θα βελτιώσει γενικά τη ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει Δεν ξέρω αν ζητάει κανεί άλλο το λόγο για το θέμα αυτό. Δεν ζητώ να ζητά κανεί άλλο το λόγο. Θα ήθελα μόνο να σα πω το εξή πώς ε, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες εβδομάδες μάλλον. Θα προετοιμάσουμε συμβαστικές προτάσεις για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για το έγγραφο αυτό. Και πιστεύω λοιπόν ότι στην επόμενη συνεδρίαση το Μάρτιο θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές. Ύστερα θα έχουμε εντολή από την Επιτροπή Γιούρη για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ποια είναι η στάση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις προτάσεις μας. Και γνωρίζουμε ασφαλώς ποιες είναι οι προτάσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υπό τη Λιτανική Προεδρία ακόμα, θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε το εργαλείο αυτό, το μέσο αυτό, προκειμένου να καταστεί λειτουργικό για τον Ευρωπαίο πολίτη, για τους ιδιώτες, για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Yes. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν συντομία, να σχολιάσω τις παρατηρήσεις που έγιναν έγινε μια συζήτηση η οποία και συνεχίζεται για το κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά κατόφλια, διαφορετικά οικονομικά όρια δηλαδή, για τους ιδιώτε και για τα νομικά πρόσωπα, για τις εταιρείε. Νομίζω ότι θα πρέπει να θυμόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε ότι η εναλλακτική για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών είναι μια εγχώρια διαδικασία όπου τα μέρη, τα μέλη θα πρέπει να ταξιδεύουν, να πηγαίνουν σε ακριάσεις, να έχουν μεγάλο κόστος. Και σε κάποια κράτη μέλη καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ε, εγγυάται την χρήση μια πιο, μιας πιο Βαρια εγχώριας διαδικασία. όταν μιλάμε για 5.000 ευρώ για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν θα το τονίσω. Κάτι άλλο. Εν συντομία. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται από απόσταση οι πληρωμές. Online. Με επιστοτική κάρτα. Αλλά προφανώς θα ήταν πιο αποδοτικό να υπάρχει μια κεντρική διαμόρφωση σε κάθε κράτος μέλος. Από το να ζητάμε από κάθε τοπικό δικαστήριο να εφαρμόσει ένα τέτοιο σύστημα. Αυτά είναι πρακτικές λεπτομέρειες τις οποίες θα πρέπει να αποφασίσουν από μόνο τους τα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να έχουν υπόψη τα ωφέλη. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Φαίνεται ότι συμφωνούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις σας. Δεν βλέπω, δεν θα κάνει άλλο το λόγο. Πολύ ωραία. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, στην ημερήσια διάταξη. Και να δώσω και να καλωσορίσω τον ε, καθηγητά Ντεπάλο και να του δώσω το λόγο για να κάνει την παρουσίασή του. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα προ όλου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερω του διοργανωτέ Μα δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την οδηγία της διαμεσολάβησης όσον αφορά εμπορικές και αστικές υποθέσεις. Πάντοτε η πύληση διαφοράς ήταν δύσκολο θέμα. Να βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται σε αυτό το μέσιο τόσο το παλιό σκίτσο. Βλέπετε ότι τσακώνεται ο ενάγων και ο εναγόμενος για την Αγελάδα και τελικά την Αγελάδα την Αρμέγιο συνήγορος. άρα επομένως η ένδικη επίλυση διαφορών είναι πρόβλημα για την ε, οικονομία και για την ενιαία αγορά, για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις. Όμως και πάλι για η δίκη είναι κάτι το οποίο στριμώνει τον κρατικό προπολογισμό σε μια δύσκολη περίοδο. Όπως ακούσατε και από τους συναδέλφους, η διαμεσολάβηση έχει πολλά πλεονεκτήματα και διευκολύνει. Και από πολύ παλιά έχει αρχίσει η χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυση διαφορών, ούτως ώστε να υπάρχει μεσολαβητής, να μην αποφασίζει αυτός για ε, τους διάδικους, αλλά αποφασίζουν εκείνοι. Αλλά αυτό είναι η διαμεσολάβηση, δηλαδή πιο φθηνή από την ενδική επίλυση διαφόρων. Και ενθαρρύνεται η διαμεσολάβηση με αυτή την οδηγία, με την οδηγία 52 του 2008 όσον αφορά κάποιες κατοχυρώσεις ποιότητας και αμεροληψίας των διαμεσολαβητών ε, όπως επίσης και για την εκτελεστότητα του αποτελέσματος της διαμεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο της Ευρώπης έκανε μια μελέτη και όμως κατέληξαν στο ότι χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση μόνο σε 0,05% των περιπτώσεων σε 27 εκατομμύρια. Δηλαδή σε... έχουμε 100.000 διαμεσολαβήσεις ενώ έχουμε 20 εκατομμύρια και άνω δίκες στα ίδια κρατημέλη, στα 27 κρατημέλη. Είναι αυτό το οποίο ορίζει το άρθρο 1. Οπότε, βλέπουμε ότι πρώτη για ένα παράδοξο. Είναι μια χρήσιμη διαδικασία, αλλά το ότι να μην χρησιμοποιείται είναι μια μεγάλη οικονομική ζημιά. Μπορεί να έχει οικονομήσει δισεκατομμύρια, όχι μόνο εκατομμύρια κάθε χρόνο. Απλώς εάν είχαμε επιτυχή κατάληξη των μισών μόνο υποθέσεων που πάνε σε δημοσιολάβηση. Άρα θα πρέπει αυτό το παράδοξο να σταματήσει. Πριν από πέντε χρόνια το δικαστήριο, το ευρωπαϊκό, ξεκαθάρισε πάρα πολύ ωραία το τι ισχύει. Αν δεν είναι υποχρεωτική, τότε δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Να ε, να είναι υποχρεωτική. Είναι κάτι το οποίο το επιτρέπει η οδηγία, αλλά δεν απαιτείται από τα κράτη-μέλη. Και μπάστος αυτό έχει να κάνει και με το κόστος. Γιατί καλή διακυβέρνηση σημαίνει ότι ο κόσμος αναγνωρίζει την αξία, αλλά δεν το χρησιμοποιεί. Να είναι σαν να λέμε για το κράνος. Τη μοτοσυκλέτα ή την ε, ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο ή τους ε, αντικαπνιστικούς κανόνες. Είναι, είπαμε, κάτι το ωφέλιμο, κάτι το λογικό, αλλά τελικά δεν επιβάλλεται το κράνος. If he could ride a motorcycle in Rome some 2000 years after his time. Οπότε υπάρχουν και οι καλές ειδήσεις. Δεν χρειάζεται να προβλέπετε υποχρεωτικά η διαμεσολάβηση. Μπορούμε. Σε αυτή τη διαδικασία να επιτρέψουμε στους διάδικους να σταματήσουν. Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός αυτοεξαίρεσης. Αυτό προέγυψε και με μια μελέτη. Είχαμε δύο ερευνητέ το 2003 που προσπάθησαν να δουν γιατί σε πολλές χώρες πόσοι είναι αυτοί που θέλουν να δωρήσουν όργανα μετά θάνατον. Ας πούμε, Αυστριακοί 100%, Γερμανοί 12%, ενώ είναι παρόμοιες οι κουλτούρες. Ποια είναι η εξήγηση, το δίπλωμα ε, οδήγησης. Επίσης, ε, έπρεπε να υπογράψουν. Πάρα πολύ λίγοι υπέγραψαν, άρα πάρα πολύ λίγοι ε, συμφώνησαν. Ή έπρεπε επίση να υπογράψουν εάν δεν συμφωνούν. Πάρα πολύ λίγοι πάλι υπέγραψαν. Αλλά αυτή τη φορά αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί ε, συμφώνησαν. Βλέπετε μέσα τι θα πει αυτό ότι σε πολλά συστήματα υπάρχει ενθάρρυνση για διαμεσολάβηση. Αλλά όταν υπάρχει κάποια διαφορά μπορούν ή να πάνε δικαστήριο ή να πάνε σε διαμεσολάβηση. Αυτό το κάνουν όλα τα κρατη τώρα. Το 2014 κάθε μια από 27 χώρες είχε λιγότερες από 10.000 διαμεσολαβήσεις και 19 από αυτές τις χώρες είχαν λιγότερα από 2.000, δηλαδή τίποτα. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα που έχει ένα σύστημα αυτοεξαίρεσης και μιλάμε για περίπου 150.000 διαμεσολαβήσεις ε, πέρσι μόλις. Και Επομένως αυτό το οποίο επιτρέπει του διαδίκου σε μερικές περιπτώσει να παραστούν σε μία ε, συνάντηση, να κοστίσει αυτό 40 ευρώ. Μετά την αρχική συζήτηση, όπου αναζητείτε μία λύση, τότε μπορεί κάποιος να αποχωρήσει χωρίς να χρειαστεί να πει τίποτα άλλο ή χωρίς να υφίσταται κάποιες άλλες ε, συνέπειες επειδή εγκατέψετε τη Μόνο εάν και οι δύο αποφασίσουν να συνεχίσουν, θα συνεχίσει τη διαμεσολάβηση. Επίση, αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι για περίπου 18 χρόνια ε, και στην Ιταλία πάρα πολύ λίγοι πηγαίνανε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, λιγότερο 5.000 και όμως εκθετική ήταν η αύξηση το 2012. Τότε που έγινε υποχρεωτική η διαμεσολάβηση το 2013 Ε, πάλι υπήρξε ε, ε, πάλι δεν μπορούσε κανείς να αποχωρήσει οπότε έπεσαν οι περιπτώσεις. Όταν υπήρξε το ελεύθερο opt-out, η, αποχώρηση ελεύθερη δηλαδή, πάλι κορυφώθηκε ο αριθμός των διαμεσολαβήσεων. Και όχι μόνο περισσότεροι πήγαν διαμεσολάβηση, αλλά και περισσότερες ήταν οι επιτυχείς καταλήξεις με αυτή την ρύθμιση της αυτοεξαίρεσης. Δεν θέλω ο να πληρώσει για, για μεσολάβηση. Λένε. Αυτό κατά 70% είναι λάθος γιατί μόλις 30% καλύπτεται. Το 70% των δικαστικών εξόδων πληρώνεται από τους υπόλοιπου. Τον υπόλοιπο λαό. Επομένως, ο λαός έχει δικαίωμα να, να ζητεί από τους διαδίκους και από τους πληρώνει τα έξοδα να δοκιμάζουν τη διαμεσολάβηση. Άρα να μην χρησιμοποιούν τα χρήματα του φορολογουμένου για τα δικαστήρια. Οι φορείς της διαμεσολάβησης στην πρώτη συνάντηση εξηγούν γιατί είναι προς το συμφέρον των διαδίκων να συνεχίσουν τη μεσολάβηση. Τώρα θα ξαναζητηθεί η οδηγία και θα εξεταστεί το που υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ας πούμε, σε περιπτώσει κοινωνικού δικαίου στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να πάνε οι διαδικοί κατευθείαν στο δικαστήριο. Θα πρέπει πρώτα απ' να δείξουν ένα σύμβουλο και όχι δημοσιολάβητη. Ε, αυτό το μελετά τώρα το, το Υπουργείο αλλά εκεί όμω δεν υπάρχει σύστημα αυτοεξαίρεσης. Ε, στην Ελλάδα επίσης ε, πάλι δεν είναι εύκολη αυτοεξαίρεση και σε επίπεδο ενωσιακό η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε κάποιες ε, νέες διατάξεις ώστε να είναι υποχρεωτική η, η διαμεσολάβηση για την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλιστικό πράκτορα και έτσι υποχρεωτικά να βρίσκεται μια λύση. Ε, αυτό βέβαια και πρόκειται να συναντήσει στεναρή αντίσταση από του επαγγελματίε. Τελικά, όχι μόνο θα είναι πιο εύκολη η ζωή του κόσμου έτσι, αλλά θα γίνει και καλύτερη αν υπάρχει μια τέτοια πολιτική που να βοηθά. Να υπάρχει δηλαδή μια τροποποίηση της οδηγίας για να χρησιμοποιήσουμε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να απαιτείται για κάποιες, κάποιες φάσεις της ε, διαδικασίας επίλης διαφόρας. Βλέπετε εδώ, τώρα τα τέσσερα στοιχεία που έχω βάλει το κόκκινο γύρω-γύρω και ε, επίσης ε, σε κάποιο σημείο θα μπορούν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσει όποιος διάδικος επιθυμεί. Να, κέντρο διαμεσολάβηση στο Αφγανιστάν. Να, να μην θεωρηθεί βλασφημία. Να, στην Καμπούλη είναι αυτό. Σας το δείχνω τώρα. Να, ένα τεστ αντοχής. Και αν ήθελε ο Θεός να ανοίξει διαμεσολάβηση, τι θα γινόταν. Θα πήγαινε ο κόσμος Ακόμα και αν ήταν ο ίδιο ο Θεό που θα έκανε τη διαμεσολάβηση. Όχι, δεν θα πήγαινε ο κόσμος, θα πήγαινε να, να μεσολαβούσε ο Θεός μόνο αν ήταν σωστό το σύστημα και οι κανόνες. Άρα όλα εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητά μα. Και σε οικογενειακό δίκαιο και σε δοραστικό δίκαιο και στο εμπορικό δίκαιο και για όλα τα κοινωνικά προβλήματα ε, θα μπορούμε να οργανωθούμε και να το καταφέρουμε Ακόμα και εδώ μέσα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Να, ποιοι αυτοί είναι οι συνεργάτες μου με τους οποίους ε, ε, ετοιμάσαμε αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Dr. Gottfried Μάσκερ, δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Αυστρίας για το τελευταίο μας ε, ζήτημα. διάβασα στο έγγραφό μου ότι συμμετείχε στην Συντακτική Επιτροπή για τη Σήμαση της Χάγης 2005 για τις Συμφωνίες Επιλογής Δικαιοδοτικού Οργάνου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα σας πω μια διαφορετική παρέμβαση. Θα μιλήσω για δύο νομικά μέσα τα οποία ισχύουν ή θα ισχύσουν σύντομα. Δεν έχω πολιτική δήλωση να κάνω. Καλούμε να παρουσιάσω δύο νομικά μέσα τη συνθήκη του 2005 της Χάγης για την επιλογή δικαστηρίου που θα τεθεί σε ισχύ στο δεύτερο ήμιση του φετινού έτους και για αναθεώρηση της κανονισμού Βρυξέλλες 1. Και τα δύο αυτά εργαλεία πραγματεύονται θέματα δικαιοδοσίας και Τη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Μιλώ για τον αντίκτυπο τώρα των δύο αυτών εργαλείων στην ε, επίλυση διαφορών σε διεθνεί συνθήκες, σε διεθνείς ε, εμπορικές συναλλαγές. Αν υπάρχει λοιπόν μια τέτοια διαφορά, κάτι θα πρέπει να γίνει. Ίσως διαμεσολάβηση, σε κάποιες περιπτώσεις όμως είναι απαραίτητο να ληφθεί μια απόφαση. Και ω εκ τούτου στην παρούσα φάση υπάρχουν δύο τρόποι να ρεθεί η απόφαση. Να απογεί απόφαση. Είτε ε, κρατικά δικαστήρια, είτε επιδιωτησία. Θα πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν τα εξή ερωτήματα. Ποιο θα αποφασίσει, ποιο κρατικό δικαστήριο, ποιο όργανο επιδιαιτησία και η απόφαση θα εφαρμοστεί στο κράτος του δικαστηρίου ή σε άλλα κράτη. Αν επιλέξει κανείς την επιδιαιτησία, θα πρέπει να ισχύσει η συνθήκη της Νέας Υόρκης, η οποία ενδεχομένως να την γνωρίζετε πιο πολύ από εσά. Πολύ επιτυχή συνθήκη. 151 κράτη έχουν προσυπογράψει. Αν υπάρξει συμφωνία επιδιαιτησία σε εμπορική έπαφη, αυτό εξαιρεί την ε, δικαιοδοσία κρατικών δικαστηρίων σε όλα τα κράτη και η απόφαση της επιδιαιτησίας θα ε, εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη που έχουν προσυπογράψει. Συνήθως λοιπόν λειτουργεί η επιδιαιτησία. Τι γίνεται όμως αν τα μέρη μια σύμβαση αποφασίσουν ότι θέλουν να εκδικαστεί σε κρατικό δικαστήριο η υπόθεσή τους. Μπορεί στην περίπτωση αυτή να συμφωνήσουν για το δικαστήριο. Να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο δικαστήριο. Να εκδικάσει την απόφασή τους, την υπόθεσή τους. Έχουμε τον παλαιό κανονισμό Βρυξέλλες 1, όπου έχει σαφείς κανονισμούς για την επιλογή ενός δικαστηρίου, όπου εξαιρούνται τα δικαστηρία άλλων κρατών μελών και η απόφαση του δικαστηρίου θα ε, εφαρμοστεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Κράτη-μέλη. Πολύ πιο λίγα δηλαδή από τα κράτη που έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη επιδετησία τη Νέα Υόρκη. Άρα το σύστημα Βρυξέλλες 1 λειτουργεί μόνο εντό τη Ένωση. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε κανόνα στι Βρυξέλλες 1 και στην παλιό και στον καινούργιο κανονισμό για την ε, επιλογή δικαστηρίου Τρίτη χώρα. Άρα δεν υπάρχει καμία νομική βεβαιότητα, ασφάλεια υπό το σύστημα των Βρυξελών 1, αν τα κράτη, αν τα διάδεκε ορίσουν το δικαστήριο ενός τρίτου κράτους ή ενός κράτους μέλους και θέλουν να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση σε τρίτο κράτος. Καμία πρόβλεψη γι' αυτό. Άρα υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κενό χάσμα νομικής βεβαιότητας. Και έχουμε λοιπόν δύο ανταγωνιστικά συστήματα, τα κρατικά δικαστήρια και την επιδιαιτησία. Αν επράτηπε μόνο για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η συνθήκη της Νέας και η Βρυξέλλες 1. Και τα δύο δίνουν νομική βεβαιότητα. Και όντω τα κρατικά δικαστήρια αποτελούν μια καλή λύση για την επιδιαιτησία. Ωστόσο, αν εμπλέκονται και τρίτα κράτη, η επιδιαιτησία δίνει νομική ασφάλεια ενώ οι σχέσεις με τρίτες χώρες δεν καλύπτονται από τις Βρυξέλλες Ένες. Άρα έχουμε μεγάλη διαφορά νομικής ασφάλειας σε σχέση με τα κρατικά δικαστήρια. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η επιλογή της συνθήκης της δικαστικής ως σκοπό θα πρέπει να έχει νομική βεβαιότητα με παράλληλο τρόπο όπως και η διαιτησία. Το παιδί εφαρμογή της συνθήκης αυτής αποκλειστική επιλογή συμφωνιών δικαστηρίων σε αστικά και εμπορικά ζητήματα, αλλά και διεθνείς υποθέσεις, δηλαδή σε εμπορικές συμβάσεις. Και ε, έχουμε εδώ τρεις βασικούς ρολ, ε, ε, κανόνες. Το επιλεγμένο δικαστήριο θα πρέπει να εκτικάσει την υπόθεση, κανένα άλλο δικαστήριο δεν μπορεί να εκδικάσει την υπόθεση και η δικαστική απόφαση του επιλεγμένου κράτους, του επιλεγμένου δικαστηρίου θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες ε, τις χώρες που έχουν προσυπογράψει. Παράλληλα δηλαδή, παράλληλη διαδικασία με την ε, συνθήκη για την Αυτό λοιπόν στα στις εφαρμογή στο δεύτερο ήμιση του έτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσυπογράψει την συνθήκη αυτή. Η αναθεώρηση λοιπόν τώρα της, ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Είχαμε δύο στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των δικαστικών συμφωνιών που λήφθησαν υπόψη στην αναθεώρηση. Καταρχάς, τώρα πια. το νέο κανονισμό Βρυξέλλες 1, Βρυξέλλες 1α, έχουμε έναν ελαφρώς διαφορετικό κανονισμό για τη συμφωνία για την επιλογή δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την ε, τεχνική αναρμόνιση με τη συνθήκη για την επιλογή δικαστηρίων. Αυτό τι σημαίνει ότι όποτε μία συμφωνία για επιλογή δικαστηρίου ισχύει σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης για την επιλογή δικαστηρίων, ισχύει και υπό τις Βρυξέλλες 1. Άρα, ω εκ τούτου είναι παράλληλη η λειτουργία τη. Δεν είναι ωστόσο αντίστοιχη και η αντίστροφη η αντιστοιχία. Οι τυπικέ ε, απαιτήσει για τη Βρυξέλλε 1 είναι, πολύ πιο, είναι κάπως πιο φιλελεύθερες. Άρα, ενδεχομένω μια επιλογή δικαστηρίου υπό τη Βρυξέλλε 1 να μην ισχύει ω ε, επιλογή δικαστηρίου υπό την συνθήκη τη Χάγη. Αλλά πάντα μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντός της ε, είναι αποτελεσματική η επιλογή αυτή. Σε τρίτες χώρες δεν είναι. Δεν ισχύει. Αλλά αν υπάρχει εγγράφος αυτή η επιλογή δικαστηρίου, ακόμα και ηλεκτρονικά, θα ισχύει και υπό τη συνθήκη και υπό τις Βρυξέλλες 1. Και υπάρχει επίσης ένας νέο κανόνας στις εκκρεμωδικίες. Υπήρξε ένα παλαιό πρόβλημα, ένα πρόβλημα παλιά με τον Βρυξέλλες 1. Υπήρξε ένας κανόνας ότι ένα δικαστήριο, αν υπάρχουν παράλληλες δικαστικές διαδικασίες σε διάφορα δικαστήρια, ε, προηγείται και το πρώτο δικαστήριο στο οποίο έγινε η αγωγή. Και θα πρέπει το δεύτερο δικαστήριο να αναστείλει τις δραστηριότητες του και να περιμένει αποτοχή της δικαιοδοσίας από το πρώτο δικαστήριο και μόνο σε περίπτωση που αποφασίσει να μην εκδικάσει το πρώτο δικαστήριο μπορεί να εκδικάσει το δεύτερο. Αυτό ακόμα και το δεύτερο δικαστήριο είχε οριστεί σε κώδικα διαντολογίας. Είναι τεράστιο πρόβλημα γιατί τα μέρη είχαν συμφωνήσει για ένα δικαστήριο και ένα από τα δύο μέρη παραβίαζε αυτή τη συμφωνία και πήγαινε σε άλλο δικαστήριο ίσως σε μια χώρα με ένα αργό διαδικαστικό σύστημα. Και έτσι μπλοκάρεται η κατάσταση και υπόθεση. Άρα, στο βρυξελλες ένα 1α, στην ε, αναθεώρηση του Βρυξέλλες 1, αναφέρεται ότι το επιλεγμένο δικαστήριο προηγείται. Ακόμα και αν το κράτος, το δικαστήριο ενός άλλου κράτους είχε δεχτεί πρώτο την υπόθεση. Και αυτό λοιπόν παράλληλα με την επιλογή δικαστηρίου, με τη συνθήκη επιλογή δικαστηρίου, γιατί στη συνθήκη επιλογή δικαστηρίου είναι σαφέ ότι το ορισμένο δικαστήριο στη συμφωνία προηγείται. Προηγείται σε σχέση με όλα τα δικαστήρια. ανταγωνιστικότητα των συστημάτων για τα κρατικά δικαστήρια. Η συνθήκη για τα επιλογή δικαστηρίων φέρνει νομική βεβαιότητα σε ό,τι αφορά την εκτίκαση υποθέσεων σε σχέση με τρίτε χώρε. Αυτό είναι καινούργιο στοιχείο. Ω τώρα, η επιλογή δικαστηρίου και η σχετική συνθήκη αποτελεί μία βιώσιμη εναλλακτική για την επιδετησία σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και αν συμμετέχουν ε, και άλλα και τρίτες χώρες. Βίβεται νομική βεβαιότητα. Αν τα κράτη, αν οι επιλέξουν μια χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη συνθήκη επιλογής ε, δικαστηρίου. Ωστόσο, όλα ε, εξαρτώνται από την επικύρωση της συνθήκης της ε, επιλογής δικαστηρίων. Αυτό θα γίνει και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και Μεξικό. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι μεγάλοι οικονομικοί φορείς θα προσυπογράψουν τη συνθήκη αυτή. Εάν το πράξουν, τότε θα υπάρχει ένα παράλληλο σύστημα με την επιδησία. Ιδάλλως, η επιτυχία της συνθήκης της Νέας Υόρκης θα μείνει απαράλλαχτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you for uh, this... Uh, σας ευχαριστούμε. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, η άποψή σας. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνουν και αυτές οι επικυρώσεις. Τώρα ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε την τελευταία μας συζήτηση για τη διαιτησία, για τη διαμεσολάβηση. Ποιος θα ήθελε το λόγο παρακαλώ. Mm. Έχω εγώ μια ερώτηση για την διαμεσολάβηση και το σύστημα opt-out. Για ε, το αστικό και το εμπορικό δίκαιο είναι εξίσου αποτελεσματικό το σύστημα ή υπάρχει κάποια διαφορά. Εγώ νομίζω ότι είναι αποτελεσματικότερο από την αλλακτική λύση. Αυτή θα ήταν μια σωστή απάντηση. Έχουμε το opt που είναι η άλλη εναλλακτική και ήρθε για 20 ε, χρόνια περίπου σε διάφορες χώρες. Το 1993 στην Ιταλία είχαν πρώτη περίπτωση διαμεσολάβησης και στη Γαλλία το 1994 και είδατε τα αποτελέσματα. Δεν λειτουργεί στο σύστημα. Αν έχετε χρόνο, ανθρωπολογικά θα σας το εξηγήσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν επιδεθείτε, δεν μπαίνω σε... διαμεσολάβηση. Αν χρησιμοποιήσετε βία, βία θα εισπράξετε. Δηλαδή, αν εγώ σας ε, ε, επιτεθώ μία φορά, θα μου επιτεθείτε τρεις. Αυτό είναι, είναι της κλιμάκωσης. Ε, δεν υπάρχει φυσική τάση, αν θες, στους ανθρώπους, στους να, να μπουν σε διαμεσολάβηση ή θα ε, παλέψουν ή θα το σκάσουν. Ε, είναι η γνωστή λέξη με έφαλο, αλλά όχι αυτή η κακή λέξη που ξέρετε όλοι που αρχίζει με F και τελειώνει με Ξέρετε ότι ένας δικηγόρος μπορεί να ε, καταφέρει να κρατήσει για πάντα μια υπόθεση. Οπότε ο στόχος μας είναι να πειραματιστούν οι άνθρωποι, όχι να υποχωρήσουν. Η Ιταλική νομοθεσία, όπως σας έλεγα προηγουμένως, δεν είναι τίποτα τελεσίδικο. Είναι μια αναπήραμα που κάνουμε μέχρι το 2017. Ε, είναι γνωστό ότι ε, υπάρχει τόσο μεγάλο βάρος και πλήθος ε, υποθέσεων που καταραίει το σύστημα μας. Δεν είναι πανάκια ούτε και ανάθυμα όμως. Θα δούμε, θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα του συστήματος. Εάν είναι θετικά, θα σταθεροποιηθεί, θα παγιοποιηθεί. Αν όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί κανείς σε καμία χώρα ε, δεν θα δεχόταν ε, τη διαμεσολάβηση αν δεν υπάρχει κίνητρο. Παραδείγματος χάρη να, τα, ε, να αφαιρείται το κόστος διαμεσολάβησης από τα δικαστικά έξω. Δεν υπάρχει τέτοια χώρα στον κόσμο που στενά δεν έχει λειτουργήσει τέτοιο σύστημα. Αν υπάρχει να μου το πείτε να μετακομίσω εκεί. Ευχαριστώ. Νομίζω φτάνουμε στο τέλος ε, του εργαστηρίου μας. Ε, σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Για μένα τουλάχιστον ήταν χρήσιμο. Ελπίζω και για σας. Ε, αφήστε που τροφοδοτεί τις εργασίες μας για τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αστικού δικαίου. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο είναι εξαιρετικά τεχνικός τομέας, νομίζω όμως πως ε, αποδείξαμε σήμερα πως υπάρχει και περιθώριο για πολιτική συζήτηση. Ελπίζω το 2017 να βρεθούμε για το επόμενο εργαστήρι. Θα περάσει πολλού χρόνο βέβαια μέχρι τότε και θα διαπιστώσουμε εάν έχει σημειωθεί ή όχι πρόοδος με την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2 θα έχουμε ολοκληρώσει τις προσπάθειες, πιστεύω, ελπίζω, μέχρι το 2017. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τους βουλευτές, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, τους υπαλλήλους που παρευρέθησαν. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε ε, για θέματα αστικού δικαίου σε ευρωπαϊκό Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερους τους εμπειρογνώμονές μας που μας διαφώτισαν και ευχαριστώ και το προσωπικό του Policy Department C, τη γραμματεία. Τόσο αναγκάστηκα να μεταφράσουν τα όσα λέγαμε. Καλό απόγευμα. Βράδυ. Καλή επάνωδο.